Colleagues, I'm very, very sorry that we, we did... Αγαπητοί συνάδελφοι, φάγαμε λίγο το χρόνο της Συνεδρίας Επιτροπής γιατί έπρεπε να συζητήσουμε κάποια θέματα μεταξύ των συντονιστών. Ήταν πολλά αυτά που είχαμε στη Μεσιαδόρια. Σας ζητώ συγγνώμη πάντως γι' αυτό και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καθίστε παρακαλώ, θα το εκτιμούσε ιδιαίτερος. Excellent. So, we need first... Τέλεια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να εγκρίνουμε το σχέδιο μερικές διάταξης. Λαμβάνω τη σιωπή σας ε, ως αποδοχή. Έχουμε και τα πρακτικά τη συνεδρίαση τη 11η Νοεμβρίου και τη συνεδρίαση τη 1η και 2η Δεκεμβρίου. Εγκρίνονται και αυτά εγκρίνονται. Κάποιες ανακοινώσεις τώρα έχω. Νομίζω ότι σήμερα η ακρόαση ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη, πάρα πολύ αποδοτική. Μας έδωσε τροφή για συζήτηση. Ήταν πηγή έμπνευση, ε, πιστεύω και για τη μεταλλωτική μα δουλειά. Θα ήθελα να ενημερώσω τους βουλευτές ότι στη γραμματεία έχουμε την κυρία Ινα Σοκόλσκα, νέο μέλος. Τη βλέπετε, έχει σηκωθεί. Ή να καλωσορίσατε Ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Η κυρία Σοκόλσκα είναι Λιθουανή υπήκος. Πριν ήταν στην Επιτροπή Γυναικών. Να τις φερθείτε καλά σας παρακαλώ. Είναι μαζί μας τώρα στην Επιτροπή τέτη. Επίσης, έχω μια άλλη ανακοίνωση για τον Παλαιγιάζ. το δεύτερο τέτοιο εγχείρημα. Γνωρίζετε ότι η πρώτη άσκηση Παλαιγιάζ ήταν μια δύσκολη συνάντηση. Περιμένω τη δεύτερη, θα την προετοιμάσουμε κατάλληλα η Γραμματεία θα επιδείξει άκρα ευαισθησία. Έχουν γίνει ήδη προπαρασκευαστικές συναντήσεις μεταξύ γραμματείας και πολιτικών ομάδων. Θα έχουμε λοιπόν τη δεύτερη άσκηση μπαλεγιάζ στην 21η Απριλίου. Έπειτα, η Bundestag θα έρθει 4 Μαΐου το μεσημέρι να επισκεφθεί την Επιτροπή μας και η μας, ο αντιπρόεδρος μας μάλλον Φραν Τίμερμαν, θα έρθει την επόμενη μέρα το πρωί, 5 Μαΐου. Μία ώρα θα καθίσει εδώ στην Επιτροπή μας. Έχετε χρόνο μπροστά σα να σκεφτείτε για να του θέσετε δύσκολα ερωτήματα και ενδιαφέροντα βέβαια ερωτήματα επί τη ευκαιρία τη επίσκεψή του στην Επιτροπή μα. Και τώρα να περάσω Το παράρτημα των σημειώσεων της Προέδρου με ποιες αναφορές θεωρούμε ότι πρέπει να ξανανοίξουν. Δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση στις πολιτικές ομάδες από αυτό, άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται οι προτάσεις. Τώρα, σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών, έχω ορισμένε ανακοινώσει. έχει διανεμηθεί ε, η μέρη διάταξη του Μαρτίου, το σχέδιο μέρη διάταξη. Το συζήτησαν οι συντονιστέ. Είπαμε ότι θα συζητήσουμε με επιταχυμένη διαδικασία τη συμφωνία TTIP, τι σχετικέ διαπραγματεύσει. Κύριο Βαλέσα θα είναι ο εισηγητή σχετική έκθεση. Το ΕΛΚ και η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έκαναν δύο αιτήματα, τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την μερίσια διάταξη του Μαρτίου. Και αν υπάρξουν και άλλα αιτήματα θα ε, προσθεθούν στις σημερινές διατάξεις και για τον Απρίλιο και τον Μάιο. Για τις εκθέσεις αποφασίσαμε να μην γνωμοδοτήσουμε για την επικουρικότητα και η ταπεινή δική μου ε, σύσταση για κάποια αμφισβητούμενα θέματα εγκρίθηκε. Uh, uh, Δεύτερο αίτημα από τους πρασίνους για επιταχυμένη διαδικασία κατεπήγοντος. Ε, δεν ελήφθη υπόψη, δεν έγινε δεκτό αυτό το αίτημα, δεν περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και συγκεκριμένα του εφετείου στην προκειμένη περίπτωση. Άρα δεν θέλαμε να προκαταλάβουμε τα πράγματα. Είχαμε επίσης ε, αιτήματα για ε, δημόσιες ακροάσεις. Είχαμε την πρόταση ECR, εκ μέρου του κ. Μαριά, ε, για να έχουμε μια δημοσία κρόαση για τι πολεμικέ επανορθώσει, η οποία όμω πρόταση δεν έγινε δεκτή. Η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ζήτησε να έχουμε μια δημόσια κρόαση για τον αντίκτυπο τη οικονομική κρίση στον τομέα τη υγεία και των φαρμάκων. Εδώ βρήκαμε μια συμβιβαστική λύση. Το τμήμα πολιτική, Policy Department, θα διοργανώσει ένα εργαστήριο με βάση έτοιμα ε, μελέτη από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ όπου θα καταγραφούν όλα τα εργαλεία και μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα αποφασίσουμε, μάλλον αποφασίσαμε ότι η κυρία Καμπεθόν Ρουή θα, έρχεται ε, σε επαφή με το τμήμα πολιτικής και θα μεταφέρει ε, στους ε, συναδέλφους εκεί τις απόψεις και τις επιθυμίες μας, ώστε να ληφθούν υπόψη. Θα πραγματοποιηθεί επίσης 26 με 28 Απριλίου σεμινάριο των Ευρωπαίων Συγχώρων του Πολίτη στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Εγώ δεν μπορώ να παραστώ, έξω και ζήτησα από όποιον ενδιαφερόμενο συνάδελφο θέλει να το κοινοποιήσει στη γραμματεία. Και αυτό μέχρι αύριο το βράδυ. Αυτές είναι οι αποφάσεις των συντονιστών λοιπόν. Ερωτήσεις υπάρχουν. Όχι. Άρα. Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Ε, συντομότατα, διότι πρέπει να προχωρήσουμε στην Επιτροπή μας, να επισημάνω και στην Επιτροπή ότι φυσικά δεν συμφωνώ με την απόφαση των συντονιστών, την πλειοψηφία τους δηλαδή, η οποία ψηφίστηκε από τον συντονιστή του ΕΛΚ και τη συντονίστρια του, του S&D να απορριφθεί η πρότασή μου για δημόσια ακρόαση για τις ε, γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις. Να ευχαριστήσω τους, ε, τις συντονίστριες της ΓΚΟΕ και του EFD που ψήφισαν υπέρ της ε, πρότασης και τις συντονίστριες των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων οι οποίες απήχαν. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσουμε να επανέλθω ξανά για το αίτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Now colleagues are waking up. Ξυπνάνε σιγά σιγά βλέπεις να αλφίσω λεδά. Ακούστε, όχι δεν θα ξαναρχίσω τη συζήτηση, δεν έχουμε χρόνο και θέλουμε να ακούσουμε και τους αναφέροντες. Να ζητήσω απλά ε, στα πρακτικά να καταγραφούν τα επιχειρήματα της ομάδας σοσιαλιστών και δημοκρατών, ε, τα οποία προανέφερα και νομίζω ότι είναι σημαντικά. Και θα διευκρινίσω και εγώ τη θέση στους υπόλοιπους ομάδας. Ε, μπορεί νομίζω να είναι διαφωτιστικό να γράφει τα πρακτικά και να καταλάβουν και οι υπόλοιποι τη θέση μας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα αυτή η πρωτοβουλία, ε, το ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το νερό είναι στη διάταξη, ναι ή όχι. Γιατί στο πρόγραμμα φαίνεται να έχει ακυρωθεί. Στη διάταξη, εν πάση φαίνεται να έχει ακυρωθεί. It is point 10 okay. on the... Είναι το σημείο 10 της ημερησίας διατάξεως, ε, διευκρινίζει η Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Okay. Did I miss anybody? No? Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Save European Citizens Initiative to end ecocide in... Λοιπόν, ε, ε, είχαμε τους EcoSide, End EcoSide in Europe, αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών τους είχαμε και στην ε, ακρόαση. Ακούσαμε ε, και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε ο οργανωτής για να μαζέψει τις απαραίτητες υπογραφές. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την ανάδραση, αυτό το feedback που έχουμε για την, προετοιμασία του κανονισμού ε, για την πρωτοβουλία των πολιτών. Η Σάχρος Μπεσέρα είναι η συγγήτρια. Ε, δεν είμαι σίγουρη βέβαια ότι είναι σωστός τίτλος αυτός που λέμε ε, η αποτυχημένη πρωτοβουλία. Δεν είναι αποτυχημένη, failed το έχουμε γράψει στα αγγλικά, αλλά ε, ε, εδώ πραγματικά με τόσες υπογραφές που μαζεύτηκαν η ευαισθητοποίηση έγινε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο σε όποιον τον ζητήσει. Νομίζω ότι η κυρία Μέρση είναι εδώ. Ναι, σας έψαχνα, δεν σας έβρισκα. Ίσως ε, μπορείτε να μας κάνετε μία σύντομη σύνοψη του περιεχομένου και του πώς έχει προχωρήσει ή θα προχωρήσει η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι, εξέχομαι μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω αυτή την παρουσίαση σήμερα εδώ. Όπως ε, ξέρετε, φαντάζομαι ότι θα έχετε λάβει και τα έγγραφα. Ε, είχαμε μία ε, πρωτοβουλία πολιτών η οποία έκλεισε στις 22 Ιανουαρίου με 114.000 14.000 υπογραφές. Ε, αποφασίσαμε πάντως να μην την κλείσουμε εν τέλει και να συνεχίσουμε να ε, μαζεύουμε υπογραφές. Είχαμε φτάσει σε 114.927 συγκεκριμένα. Αποφασίσαμε λοιπόν να συνεχίσουμε την συλλογή υπογραφών γιατί πιστεύουμε ότι είναι ακόμα πολλοί οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν και να προσυπογράψουν αυτήν την ε, πρωτοβουλία. Ε, ήδη ε, από τις 22 Ιανουαρίου μέχρι, του 14 μέχρι τώρα έχουν μαζευτεί ακόμα 70.000 υπογραφές ε, και επομένως έχουμε ένα σύνολο 185.000 ε, πολιτών που στηρίζουν ε, αυτήν την πρόταση. Θα ήθελα να σας εξηγήσω εν συντομία λίγο αυτά που περιλαμβάνει η πρωτοβουλία. Η κυρίαρχη ιδέα είναι πάρα πολύ απλή, δηλαδή ε, ότι η ευρεία κλίμακος περιβαλλοντική καταστροφή θα πρέπει να θεωρείται έγκλημα. Ένα έγκλημα το οποίο, ε, για το οποίο θα πρέπει να είναι υπόλογη ε, ή ε, αυτοί που έχουν πάρει αποφάσεις. Κάποιος θα πρέπει, σε κάποιον θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Αλλά βεβαίως εδώ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις, στους υπευθύνους και τα χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα τα οποία τα οποία έχουν χρηματοδοτήσει αυτού του είδους τα προγράμματα. Η ιδέα δεν είναι καινούρια, συζητιέται εδώ και 50 χρόνια ε, και μάλιστα η, αυτή η οικολογική καταστροφή συμπεριλήφθηκε ε, σε, ένα, ε, σε έναν κατάλογο ο οποίος αφορούσε όλα τα εγκλήματα κατά της κατά της ειρήνης μαζί με την γενοκτονία, μαζί με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μιλάμε επομένως για ενέργειες οι οποίες γίνονται ήθελημένα και με σκοπό την καταστροφή. Θεωρούμε λοιπόν ότι η οικολογική καταστροφή πρέπει να θεωρείται ε, έγκλημα. Ε, καταρχήν ε, θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί, ήταν η ιδέα να συμπεριληφθεί και στην συνθήκη της Ρώμης. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή υπάρχει το άρθρο 8.2b, ε, ε, το οποίο ε, εδάφιο 4, το οποίο εξακολουθεί να κάνει αναφορά σε ευρεία κλίμακας και μεγάλη σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον. Και αυτό θεωρείται, θεωρείται έγκλημα πολέμου. ο νόμος ε, καταδεικνύεται ότι μπορεί να λειτουργήσει και έχει λειτουργήσει πολλές φορές, αλλά εν τέλει αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση έτσι ώστε να ισχύσει ο νόμος τι είναι ακριβώς αυτή η οικολογική καταστροφή. Βλέπετε εδώ ε, διάφορους ορισμούς. Ε, είναι η διευρυμένη, η μεγάλη ε, καταστροφή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό πρόβλημα σε μεγάλη περιοχή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τα οικοσυστήματα ε, και όχι γενικά και όχι μονάχα την καταστροφή ενός συγκεκριμένου είδους ε, ε, γιατί το ένα πράγμα μπορεί να είναι συνδεδεμένο με κάτι άλλο και επομένως να υπάρχει μια αλυσίδα αλληλεπιδράσεων. Ε, είναι γεγονός ότι σε μερικές ε, περιπτώσεις ε, μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη καταστροφή στους ανθρώπους ή σε άλλα είδη τα οποία παρεπιδημούν στην περιοχή. Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε μείωση ή διαφοροποίηση ή ταραχή της καλής διαβίωσης όλων των εμβίων όντων σε μια περιοχή μπορεί να θεωρηθεί οικολογική καταστροφή τροφί Ε, Πολλές ε, είναι και οι ε, καταστροφές οι οποίες γίνονται όχι μονάχα στην ε, Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες ας πούμε στις καναδικές στη, καναδική επικράτεια στους αμολόφους ή επίσης στην, στον Αμαζόνιο. Μπορεί κανείς επίσης να δει και την κατάσταση στη Ρουμανία, στην περιοχή Ρώσια, Μοντάνα ή ακόμα και τα ε, τα, τα κοιτάσματα χρυσού και τις εξορίξεις τους στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, ε, καθώς επίσης ε, και τις απειλούμενες εξορίξεις που μπορεί να γίνουν στα Κανάρια νησιά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθούν πλέον τα σωστά εργαλεία και βεβαίως η οδηγία, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Οικολογική Καταστροφή θα μπορούσε να είναι ένα από τα εργαλεία αυτά. Να βρεθούν, λέω, τα σωστά εργαλεία έτσι ώστε να μπορέσουν οι ίδιες οι κοινωνίες να αντιταχθούν και σε αυτή την καταστροφή και να προστατέψουν τις περιοχές τους. Ε, Βεβαίως ε, η Ευρωπαϊκή Ενωσιακή Νομοθεσία μπορεί να καλύψει μέσω της οδηγίας αυτής ε, τις καταστροφές οι οποίες γίνονται στην ε, ενωσιακή επικράτεια εάν έχουν γίνει από Ευρωπαίους πολίτες και αν έχουν γίνει από εταιρείες οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στην ενωσιακή επικράτεια. Εάν οι εταιρείε αυτές εισάγουν ή εξάγουν αντίστοιχα προϊόντα τα οποία σχετίζονται ή ακόμα χρηματοδοτούν αυτές τις ε, ε, διαδικασίες. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την δικαιοδοσία ε, έτσι ώστε να κάνει τέτοιου είδους νομικά κείμενα. Και η αρμοδιότητα αυτή έχει επιβεβαιωθεί πρώτα απ' όλα μέσω της καταγραφής και καταχώρησης της πρωτοβουλίας των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπέρανε ότι όντως μπορεί να προταθεί αυτό το νομοθέτημα. Δεύτερον, ε, πολλοί είναι οι νομικοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι ε, έχουν αναφερθεί στην Οδηγία 2008-99 για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει νομικά ή μάλλον να νομοθετήσει όσον αφορά τα θέματα αυτά. Ε, λέγαμε λοιπόν ότι η οικολογική καταστροφή μπορεί να ε, δώσει μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη, μπορεί να συμβάλλει εις την δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος και επομένως να αυξήσει την ευζοία, το ποσοστό ευζοία στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ε, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία όμως θα καλύπτονται από το νομικό σύστημα. Το ισχύον νομικό σύστημα ε, οδηγεί ε, σε μια κατάσταση όπου το κέρδος είναι αυτό το οποίο έχει, παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Οποιοςδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει φιλική προς το περιβάλλον ε, διαδικασία ε, θα πρέπει να πληρώσει περισσότερο. Αυτό όμως ε, δεν είναι καθόλου θετικό. Αυτοί οι 185.000 άνθρωποι οι οποίοι προσυπέγραψαν την πρωτοβουλία πιστεύουν ότι θα πρέπει να δοθούν πλήρες δυνατότητες έτσι ώστε να έχουμε πρόληψη από τις οικολογικές καταστροφές. Ε, θα πρέπει να υπάρξει αυτό το εργαλείο για το τέλος της οικολογικής καταστροφής ε, γιατί μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη και μπορεί να αποβεί υπέρ των πολιτών. Έχουμε 185.000 λοιπόν πολίτες από όλη την Ευρώπη και το βλέπετε σε αυτό το γράφημα τις ηλεκτρονικές μόνο υπογραφές βλέπετε. Θα ήταν πολύ πιο πολύπλοκο να σας δώσουμε και στατιστικά στοιχεία για όσους πέρασαν ε, σε, έντυπο, σε έντυπα μέσα. Ε, βλέπετε λοιπόν ποιοι ε, ουσιαστικά ψηφίζουν πέρα αυτής της πρωτοβουλίας πολιτών. Είναι από πολλές διαφορετικές χώρες, άρα συσπηρώσαμε τον κόσμο και όλοι συμμερίζονται την άποψη ότι έχει ισχύ ο, νόμο και αυτό, ο νόμος για να αλλάξει η οικονομία, να στραφούμε μακριά από τον άνθρακα και να βοηθήσουμε τι μελλοντικέ γενιέ να ζήσουν καλύτερα. Θα πρέπει και μπορεί η Ευρώπη να οδηγήσει. Όπω ακούσαμε το πρωί, υπήρχαν πολλά προβλήματα με διάφορε πρωτοβουλίε πολιτών. Χάσαμε πολλέ υπογραφέ και εμεί. Πρέπει να σα πω ότι με βάση τα δικά μας στατιστικά στοιχεία, Μπορεί να μην είναι 100% ακριβή βέβαια γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε όλα τα ε, δεδομένα γιατί τα έχουν οι περισσότερες κομισιόν. Με βάση τα δικά μας στοιχεία χάσαμε το 44% ε, των ε, ανθρώπων, δηλαδή μόνο το 44% από αυτούς που τα υπέγραφαν υπέγραψαν. Και ποια ήταν η εξήγηση που μας έδωσαν ότι χάθηκαν στα συστήματα συλλογής υπογραφών online ότι δηλαδή είναι πολύπλοκο, έχει πολλά τετραγωνίδια, αν κάνεις κάτι λάθος δεν σου βγάζει κάτι κόκκινο, σου ξαναβγάζει την οθόνη, ε, δεν μπορείς να το καταλάβεις ότι κάνεις λάθος. Ε. Και επειδή ποτέ δεν λαμβάνεις την επιβεβαίωση, ε, όπως έλεγε και μία συμμετέχουσα σήμερα το πρωί, δεν ήξερε καν για ποια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία έχει υπογράψει. Ε, πρέπει λοιπόν, ε, αφού έχουν συμπληρώσει, να βάλουν ε, submit, υποβολή δηλαδή, αλλά μπορεί να του ξαναγυρίσει στην ίδια σελίδα. Και δεν έχουν καταλάβει αν έκαναν κάτι λάθο ή αν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Χάσαμε πολλέ υπογραφέ με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά ήταν επιτυχημένη η προσπάθειά μα γιατί καταφέραμε να συγκροτήσουμε μια ομάδα. Ε, Όπω είπα, συγκεντρώσαμε πολλέ υπογραφέ, κερδίσαμε την υποστήριξη οργανώσεων, ομάδων και όπως προείπα, ουσιαστικά είμαστε η μόνη πραγματικά ε, πρωτοβουλία πολιτών. Δεν έχουμε πίσω μας κάποια οργάνωση, είμαστε απλά μια ομάδα πολιτών, οι οποίοι συσπηρωθήκαμε πίσω από αυτό το στόχο. Ε, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο προς το παρόν, δεν υπήρχε κάποια δομή προηγουμένως. Επομένως για μας σίγουρα ήταν πολύ πιο δύσκολο, εξού και είμαστε και πολύ υπερήφανοι που συγκεντρώσαμε 185.000 υπογραφές. In Europe... Στην Ευρώπη έχουμε το προνόμιο της ελευθερίας, ε, της έκφρασης, συμμετέχουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες και πιστεύουμε ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε, να ε, διαμορφώσουμε το μέλλον. Και αυτό μας ενέπνευσε να αναλάβουμε αυτή την τεράστια πρόκληση, χωρίς ε, ουραντική δομή, χωρίς εμπειρία, χωρίς χρηματοδότηση. Επειδή όλοι πιστεύουμε ότι αν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος με το status quo, αντί να παραπονείται πρέπει να αναλάβει δράση, να προτείνει εναλλακτικέ λύσεις. Και ένα νόμο για την οικολογική καταστροφή είναι μια τέτοια λύση. Έχουμε στην Ευρώπη την τεχνολογία, τη δυνατότητα να ηγηθούμε. Έτσι θα μειώσουμε και τι εκπομπές, αλλά θα ε, ανεξαρτητοποιηθούμε και από του ανατολικού γείτονε. Οι ηγέτε μας πρέπει να κάνουν αυτό το ποιοτικό ε, άλμα ε, και όλοι εδώ που είστε σήμερα παρόντες πρέπει να βοηθήσετε να το κάνουμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Όπως γνωρίζετε, Ω εργαλείο αυτή η πρωτοβουλία πολιτών αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, έξω και είναι και εξωσημείωτο που έδωσαν τα προσωπικά του δεδομένα 185.000 πολίτες για να στηρίξουν αυτόν τον προτινόμενο νόμο. Σας παρακαλώ λοιπόν και εκ μέρου των μελλοντικών γενεών να φροντίσετε ε, να συνεχιστεί ο διάλογος των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, αλλά όχι μόνο αυτό. Αυτός ο διάλογος να οδηγήσει και σε μια πραγματική έκβαση που θα σημαίνει ε, την ψήφιση ενός νόμου που θα προστατεύει και τα ε, οικοσύστημα της Ευρώπης και τα οικοσύστημα όλου του κόσμου. Ευχαριστώ. Thank you very much and thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που πέρασες όλη αυτή την ημέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω πως είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Τώρα με μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο στην Όλγα Κούρπιτς. Νομίζω είναι παρούσα. Ίσως ε, νομίζω στον κύριο Χάνσο Πάτα που ξέρει την ουσία του θέματος. Βεβαίως, ο λόγος είναι δικό σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, της ε, ευχαριστίας μας για αυτή την πρόταση που έκαναν ε, για την δράση αυτή και για την προσπάθεια της προστασίας των οικοσυστημάτων από την καταστροφή και την απώλεια. Βεβαίως και μοιραζόμαστε τα, τους στόχους αυτούς της πρωτοβουλίας γιατί χάνονται πάρα πολλά οικοσυστήματα. Η βιοπικιλότητα κινδυνεύει παγκόσμια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να υπογραμμίσουμε τη δυσκολία που δημιουργούν τα θέματα αυτά στις ε, πολίτες μας και πόσο πολύ πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με σοβαρό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία 50 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο πλέγμα περιβαλλοντικού δικαίου έτσι ώστε να διατηρήσει την, φυσική της κληρονομιά, να αντιμετωπίσει την αλλαγή του κλίματος και αυτό το κάνω απαριθμώντας κάποιους από τους πιο σημαντικούς κλάδους που αφορούν αυτή την αναφορά. Αναγνωρίζουμε πως η νομοθεσία από μόνη της δεν εξασφαλίζει πως θα πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Θα χρειαστεί να εφαρμοστούν όλα αυτά μέσω της ανθρώπινης δράσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν μέσα, εργαλεία, μεθόδους. Έχουμε στην Ευρώπη τα απαραίτητα. Και αυτό αναφέρεται και από την πρωτοβουλία αυτή, αλλά δεν είναι πάντα ε, αποδοτικά. Εμείς είπαμε πως πρέπει να μετακινηθούμε από τη δημιουργία νέων νομικών κανόνων στην αξιολόγηση των υφισταμένων και στην καλύτερη λειτουργία αυτών που ήδη υπάρχουν να αναφερθώ σε δύο μέσα τα οποία είναι μεγάλη σημασία για τον κλάδο που καλύπτει αυτή η πρωτοβουλία. Είναι η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη και για το ε, περιβαλλοντικό έγκλημα. Είναι η 99 του 2008 και έχουμε και το θέμα τη προστασία του περιβάλλοντο από εγκληματικέ δράσει. Δηλαδή, σοβαρέ παραβιάσει του περιβαλλοντολογικού δικαιού τιμωρούνται με αναλογικά και αποτρεπτικά ε, ποινικά, ε, ποινικές ποινές. Δηλαδή, ό,τι προκαλεί θάνατο, μεγάλη ζημία, αναπηρία στην, ε, στους ανθρώπους, στα ζώα, στα φυτά, στον ατμοσφαιρικό αέρα και στα ύδατα. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει αυτή η μεγάλη καταστροφή των οικοσυστημάτων ε, να καλύπτεται γιατί είναι στα πλαίσια αυτής της νομοθεσίας που εφαρμόζεται για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος στην ε, Ευρώπη. Έχουμε και την 34 ε, του 2005 για την περιβαλλοντική ευθύνη, για την πρόληψη και για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών η οδηγία αυτή είχε σκοπό να προλάβει τις άμεσες απειλές προς το περιβάλλον, στο να αποκαταστήσει το περιβάλλον ε, και να εξασφαλίσει τη βιοποικιλότητα ε, και να διατηρήσει τα ύδατα και τα εδάφη. Εκεί υπάρχει πολύ ε, καθαρά περιγραφόμενη ευθύνη που βαραίνει τους εμπορευόμενους και τους εμπλεκόμενους οι οποίοι μετά είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν το φυσικό πόρο στην κατάσταση που ήταν πριν την ε, βλάβη και να αναλάβει και όλο το κόστος αυτής της αποκατάστασης. Αυτά λοιπόν ε, είναι πολύ σχετικά με τα όσα θέματα έθεξε αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών στην Ευρώπη και στα πλαίσια μια μελλοντική οδηγία θα λυθούν διόντω υπόψη. Η υπερβολική οδηγία για την ευθύνη, την παραγωγική ευθύνη αυτή τη στιγμή περνάει από αναθεώρηση, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την συνεκτική προσέγγιση και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Βασίστε αυτό στην εμπειρία που έχουμε αποκτήσει με την οδηγία αυτή και πώς εφαρμόστηκε από όλα τα κράτη-μέλη και έχουμε εντοπίσει τις προκλήσεις και τις ελλείψεις που έχουμε στην εφαρμογή για να τη βελτιώσουμε. And let me conclude by uh, stressing the fact that citizens undoubtedly Να σας πω πως η πρωτοβουλία των πολιτών έπαιξε ένα πολύ κρίσιμο ρόλο. Για, θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει το ρόλο αυτό για να εξασφαλίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος στα κράτη-μέλη. Αυτή η πρωτοβουλία πολιτών λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστεί με τους δικού μας στόχους που είναι η καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα και όπου αυτό το προσφέρει η ευρωπαϊκή, ε, το προσφέρουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες ε, που προστατεύουν το περιβάλλον γιατί έχουμε πολλές οδηγίες και μία από αυτές είναι η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη. Και αυτό σας το είπα για να σας πω, ε, σας δώσω κάποια παραδείγματα, όπου γίνονται εκεί κάποιες περιβαλλοντικές μελέτες σκοπιμότητας και όπου ορίζεται πως οι πολίτες οι οποίοι επηρεάζονται από τις βλάβες ή οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα πρέπει να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές έτσι ώστε να ανοιχνευτεί η δυνατότητα βλάβη βλάβης ζημίας και να ληφθεί μετά η ενδεδειγμένη τράση. Υπάρχουν και κάποιες μη νομοθετικές πράξεις, για παράδειγμα αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην ε, στρατηγική μας για το 2020 και τα θέματα της συμβολής της ε, ε, πράσινης ανάπτυξης στη γεωργία ε, στην κτηνοτροφία και στην ε, στρατηγική, στη δασική μας στρατηγική. Υπάρχει ανάγκη να κάνουμε πρόοδο. Και θα πρέπει αυτό να γίνει σε διάφορα κεφάλαια, έτσι ώστε να πάψει πια η καταστροφή του οικοσυστήματός μας και οι μελλοντικέ γενιές να μπορούν να ζήσουν μέσα σε ένα ε, βιώσιμο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much. Εμείς σας ευχαριστούμε. Αυτή ήταν νομίζω η συμβολή της Κομισιόν στη συζήτηση και τώρα οι συνάδελφοί από την Επιτροπή μας έχουν το λόγο. Ο κύριος Τέιλορ θα ξεκινήσει, η κυρία Ντανόκα στη συνέχεια. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας για την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε τη διαδικασία αυτή αποτυχία ε, ούτε και στην προκειμένη περίπτωση που δεν συγκέντρωσε αυτή η πρόταση ένα εκατομμύριο υπογραφών. Το θέμα είναι ότι ευαισθητοποιήθηκε η κοινή γνώμη. Και το ίδιο ισχύει και για όλες τις άλλες ε, πρωτοβουλίες που δεν γίνονται δεκτές. Η Κομισιόν ε, αναγνωρίζει την ανάγκη νομοθεσίας για την οικολογική καταστροφή. Τα είπε άλλωστε όλα η αναφέρουσα. Και εγώ θεωρώ ότι έχουμε και εμείς ευθύνη μια τέτοια δέσμη προτάσεων να, να πάρει ε, ορμή, να έχει όθηση, να αναγνωριστεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να τελματωθεί ε, εδώ η προσπάθεια να σταματήσει. Καλό λοιπόν την Επιτροπή μας ε, να συστήσει συζήτηση, ίσως επίπεδο λομέλες κατά κάποιο τρόπο, της πρωτοβουλίας τέλος στην οικολογική καταστροφή, με συνεργασία Επιτροπών ΕΝΒΙ ΛΥΜΠΕ. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω η Επιτροπή ΠΕΤΗ να διεξαγάγει, να αναθέσει την εξαγωγή μιας ανεξάρτητης μελέτης για ένα νόμο περί τέλους ε, της οικολογικής ε, καταστροφής. Χαιρετίζω τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, δεν ξέρω πόσες ε, καταγγελίες και διώξεις έχουν γίνει με βάση το ποινικό δίκαιο, αλλά είναι σημαντικό και είναι και η πεμπτουσία του όλου ζητήματος να υπάρχει ε, μία γραμμή ευθύνης, ε, να οριστούν αυτές οι αξιόπινες πράξεις και να επιβάλλονται και ποινές για την τέλεσή τους. Ένας τέτοιος νόμος ε, θα μπορούσε να δώσει σάρκα και οστά στην αρχή της προφύλαξης, της αρχής ορυπαίνων πληρώνει. Και μια ιδέα που πρέπει πλέον πιστεύω να γεννηθεί, αφού κυοφόρησε για πολύ καιρό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος τώρα, η κυρία Ντανόκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα. Έχω ένα ερώτημα για τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσαμε τα επιχειρηματά σας. Είπατε, αν κατάλαβα καλά τουλάχιστον, ότι υπάρχει αρκετή νομοθεσία, μιλήσατε για τις φτάμενες οδηγίες. Άρα, ποια θα ήταν η απάντησή σας αν είχαν συγκεντρωθεί οι ε, ένα εκατομμύριο υπογραφέ. Θα αλλάζατε θέση ή όχι. Η απουσία των περίπου 800.000 υπογραφών σας δίνει το δικαίωμα πολύ απλά να αγνοήσετε αυτή την πρωτοβουλία πολιτών. θα μπορούσατε να πάρετε ένα χαρτί ε, σαν και αυτό στα χέρια σας, να κάνετε κάποιες αλλαγές και να προτείνετε μια σχετική οδηγία, έστω και αν έχει συγκεντρώσει μόνο 185.000 υπογραφές αυτό το έγγραφο. Αλλά ε, δεν σας καταλαβαίνω πολύ καλά. Τα προβλήματα τα βλέπετε, τα κενά τα βλέπετε. Η αντίδρασή σας ποια θα ήταν, αν υπήρχε αυτό το 1 εκατομμύριο υπογραφών. Το πρωί δυστυχώς δεν πάρει στην ακρόαση. Νομίζω παρουσιάσατε και εκεί την υπόθεσή σας για δεύτερη φορά. Στον σας τρέφομαι. Πώς να το πω τώρα. Ποιο κράτος θα αρμόδιο για την ε, συγκέντρωση των ηλεκτρονικών υπογραφών, γιατί από ό,τι ξέρω πρέπει να καταχωρήσετε ε, σε ένα κράτος την ε, ιστοσελίδα που θα έχετε δημιουργήσει για τη συλλογή αυτών των υπογραφών. Μήπω δεν κάνατε την καλή επιλογή, μήπως επιλέξετε λάθο κράτο. Ε, κάτι τέτοιο θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Mrs. Βαλίνα. Κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ. Πρέπει να συγχαρούμε καταρχάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και την Επιτροπή μας η οποία ακούει, υποδέχεται τους ε, ανθρώπους οι οποίοι προωθούν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών που δεν συγκέντρωσαν τον εκατομμύριο. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε χώρες όπως η δική μου, την Ισπανία, όπου 12 νομοθετικές πρωτοβουλίες, λαϊκές πρωτοβουλίες που είχα συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 500.000 υπογραφές, δεν ε, πήραν το πράσινο φως και θα ήθελα να πω ότι πρέπει να συγχαρούμε τους ε, αναφέροντες που πρόωθησαν αυτή την πρωτοβουλία. Αυτές οι αναφορές ε, είναι θα έλεγα και η πλειοψηφία, ε, δηλαδή αναφορές που εξετάζουμε στην πλειοψηφία τους έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, τη φύση. Έχουμε το δίκτυο Natura, προστατευόμενες περιοχές, ε, στην Αλμερία έχουμε μια περίπτωση εκεί με εντατική καλλιέργεια, βιομηχανική Δύο εκατομμύρια και ένα εκατομμύρια ελιά που ε, φυτεύονται, μειώνει το υδροφόρο ορίζοντα. Όταν είχαμε 70 λίτρα το δευτερόλεπτο, το έχουμε 3,4 ή 4 λίτρα ανά δευτερόλεπτο. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε τη φύση, το περιβάλλον, Επομένως σας συγχαίρω και ελπίζω η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει πιο σοβαρά από ό,τι μέχρι τώρα τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Mrs. Ε, thank you. Ε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους αγωνίζονται για αυτή την πρωτοβουλία για την οικολογική καταστροφή είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσετε την πίεση έτσι ώστε να υπάρξει νομοθεσία επ' αυτού. Εντόνως ε, υποστηρίζω την ε, έκκληση για δράση που απευθύνατε προς τους ε, βουλευτές και που επανέλαβε και ο Keith Taylor προς τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υπάρχει ίσως και κάποια άλλη επιτροπή στην οποία θα μπορούσαμε να στείλουμε αυτήν την πρωτοβουλία. Δηλαδή να μην την αφήσουμε μονάχα στην ΕΜΒ και στη ΛΥΜΠΕ, αλλά και στην Άγκρη, στην Επιτροπή που ασχολείται με τη Γεωργία και την, ε, και τα, την Αλληλεία, γιατί ξέρουμε ότι πολύ συχνά οι αποφάσεις για την ε, αλλιευτική πολιτική, την γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Προκαλεί δηλαδή καμιά φορά η κοκτονία η ίδια. Οι ευρωπαϊκές ε, πολιτικές και η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και, αυτό, και αυτή την πτυχή του θέματος. Από τη μία έχουμε ε, την ε, ε, κοινή γεωργική πολιτική η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στην ανάπτυξη και όλο και περισσότερη ανάπτυξη και από την άλλη πλευρά ξεχνούμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματά μας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Άλλη μια συνάδελφος, η Ελεονόρα και μετά θα πρέπει να κλείσει ο κατάλογος των αγορητών και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ελεονόρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσίαση που μας κάνατε, αλλά και για την προσπάθεια που έχετε καταβάλει για να συλλέξετε όλες αυτές τις ε, υπογραφές και να ε, διεξάγετε αυτόν τον αγώνα, γιατί πρόκειται για πραγματική μάχη. Βεβαίω όλα αυτά ε, είναι πολύ σωστά που λέτε. Βεβαίως ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί ε, σωστά ο ευρωπαϊκός κανονισμό και αυτός θα έπρεπε να είναι ιδεοδό ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου βλέπουμε να υπάρχουν παραβιάσεις το, της νομοθεσίας ή περιπτώσεις εσφαλμένης ή ελλειπούς ε, η εφαρμογή ε, Θα πρέπει επίσης ε, να γίνουν μελέτες στα κράτη-μέλη. Ίσως υπάρχουν και ήδη μελέτες στα κράτη-μέλη, επιδημιολογικές και λοιπές, που μπορούν να μας βοηθήσουν να περιγράψουμε σαφέστερα τα διάφορα προβλήματα τα οποία προκαλούνται από την μόλυνση, από τις, τα φέσα απορριμμάτων, από μια σειρά στοιχεία τα οποία μπορεί να, είναι, να έχουν πραγματικά πολύ κακό αποτέλεσμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επιστημονικές αναλύσεις του αέρα, του εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα και ε, τα συμπεράσματα να γίνονται γνωστά, να δημοσιοποιούνται έτσι ώστε να τα ξέρουν και οι πολίτες γιατί ε, όλοι ζούμε στο ίδιο, στην ίδια Ήπειρο και επομένως πρέπει να μοιραζόμαστε ε, τους ίδιους προβληματισμούς. Όσον αφορά τώρα αυτά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα βλέπουμε ότι το Νοέμβριο του 2014 η Eurojust αναφέρει στην τελευταία της έκθεση ε, το γεγονός ότι πολύ συχνά έχουμε περιβαλλοντικές παραβιάσεις οι οποίες παραμένουν ατιμόρητες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβουμε δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα τα οποία τελικά έχουν απόλυτο αντίκτυπο σε όλες τις χώρες μέλη. Ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Θέλετε να πάρετε το λόγο για να δώσετε μια πολύ σύντομη απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω σύντομα από τη θεσμικής πλευράς στην κυρία Ντανόκα. Η ερώτησή σας είναι υποθετική βέβαια. Στο πρώτο τμήμα του hearing ε, όσοι ήταν παρόντες θα διαπίστωσαν ότι εμείς ε, θέλουμε να έχουμε input πολλών ε, ιδεών ε, και βεβαίως η Κομισιόν μετά έχει πρωτοβουλία κινήσεων, αλλά η Κομισιόν αναλαμβάνει πρωτοβουλία παίρνοντας ερεθίσματα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και νομίζω ότι ο Επίτροπος σε αποσαφήνισε σήμερα το πρωί ότι ε, ενδεχομένως αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν ε, έφτασε, δεν κατάφερε να, να περάσει το, ε, τον αριθμό των απαιτουμένων υπογραφών αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντική. Ξέρουμε ότι ο κανονισμός ε, για την πρωτοβουλία των πολιτών έχει λόγο που υπάρχει ε, και διευθετούνται εντός αυτού όλες οι διαδικασίες ε, και πρέπει να σας πω ότι και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τις πολιτικές και τις αποφάσεις που παίρνει η Κομισιόν σαν κολέγιο που λαμβάνεται από ορισμένους, ας πούμε, από μικρό αριθμό ε, τι θα, ε, εδώ αναρωτιόμαστε τι θα γινόταν αν είχαμε φτάσει αυτό το ένα εκατομμύριο ε, υπογραφών. Είναι τελείως διαφορετικό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και μαζί μας, που μας δώσατε αυτή την ειλικρινή απάντηση. Και βεβαίως είναι καλό να συνεργάζονται τα θεσμικά όργανα σε τέτοιου είδου πρωτοβουλίε. Πολύ ωραία. Ακούσαμε τις δυσκολίες σας, κυρία Μέρτσα, μας είπατε τις δυσκολίες της συλλογή υπογραφών και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά που ακούσαμε, θα πρέπει να, ακούσουμε την, ε, να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία την οποία έχουμε συλλέξει από όσα μας έχετε πει ε, και ε, περνάμε λοιπόν στην Μπεατρίς Μπεσέρα η οποία είναι η συγγήτρια για το θέμα του κανονισμού της πρωτοβουλίας των πολιτών. Λοιπόν, θα μπορούσαμε λοιπόν να λάβουμε γνώση ε, όλων αυτών που ακούσαμε ε, και να στείλουμε όπως ε, ακούστηκε ε, το θέμα αυτό να το προωθήσουμε και στην ΕΜΒΗ και στην ΛΥΜΠΕ αλλά επίσης και στην Επιτροπή Γεωργίας αλλά και Αλίας. Φαντάζομαι ότι δια της σιωπής σε αυτά που μόλις είπα και επομένως μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Η κυρία Μίτσι πρέπει να φύγει γρήγορα για την Μάλτα και επομένως θα δώσω τον λόγο στην Περατρίς πρώτα και μετά αμέσως σε εσάς κυρία μου. Θα ήθελα για τη γνωμηδίτηση που θα γίνει αυτή για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των πολιτών. Πρέπει να σας πω πως παρόλο που ήμασταν όλοι και το πρωί στη συνεδρίαση, είναι σημαντικό να πούμε πως συνέβη αυτή η συνεδρίαση η οποία όχι μόνο μας φώτισε, αλλά μας επέτρεψε να ανταλλάξουμε πληροφορίες οι οποίες συγκλίνουν όλες προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, έχουμε όλη την εντύπωση και όλοι έχουμε μια κοινή άποψη πως για αυτές τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες των πολιτών πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα. Να ξεπεράσουμε τους φραγμούς, να αφαιρέσουμε εμπόδια. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι πραγματικά χρήσιμες. Καρποφόρες να είναι πρωτοβουλίες των πολιτών καταρχήν, αλλά ευρωπαϊκές, έτσι ώστε να έχουν σημασία για τον Ευρωπαίο πολίτη. Διδάγματα από τα όσα πετύχαμε με τις πρωτοβουλίες που έφτασαν όλες τις υποχρεώσεις και με αυτές που δεν τα κατάφεραν και εμπειρία από άλλους οργανισμούς που έχουν συμμετοχή πολιτών, έτσι ώστε με τα εργαλεία αυτά να φέρουμε την αλλαγή. Το είπαμε σήμερα το πρωί γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα συνεισφοράς και των πανεπιστημίων με την έκθεση, με την γνωμοδότηση που έχουμε μπροστά μας για την έκθεση της ΑΦΚΟ θα έχουμε την ευκαιρία όχι μόνο να συνεργαστούμε γιατί είναι κοινή η άποψή μας και συμπίπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και αντίθετα με τόσα συμβαίνει με άλλες γνωμοδοτήσεις, θα είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα προωθήσει αυτή η γνωμοδότηση είναι η λήψη αποφάσεων και δράσεων που θα είναι αποτελεσματικές για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που συμπεριλαμβάνονται και τα οποία νομίζω αρχικά μας βρίσκουν σύμφωνος. Δηλαδή, Υπάρχει αυτή η ενιαία θηρίδα, για να τη χαρακτηρίσω έτσι, σε όλα τα κράτη-μέλη που μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή Επιτροπή Αναφορών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε και αυτή την πρωτοβουλία αλλά και τις πληροφορίες που συνδυάζονται με αυτήν. Υπάρχουν θεσμοί, υποδομές, προσωπικό. Μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να ξέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες σε ποιον πρέπει να αποτανθούν. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα πρόσβασης, για παράδειγμα, στο να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία. Δηλαδή, θα πρέπει να μπορεί κανείς να ε, εντοπίζει με τον ίδιο τρόπο τους υπογράφοντες. Αυτό είναι ένα θέμα, η ενιαία ευρωπαϊκή ταυτοποίηση του υπογράφοντα. Αυτό μένει να γίνει, όπως επίσης και να εξασφαλίσουμε όχι μόνο την νομική κάλυψη όσων προωθούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, αλλά και την νομική αρρωγή που μπορεί να τους προσφερθεί. Θέλουμε να συστρατευτούμε περισσότερο, να είναι διάφανη διαδικασία και να εξασφαλίσουμε πως γίνεται γνωστή. Ξέρουν οι πολίτες αλλά και όσοι προωθούν τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλίες πως υπάρχουμε Δηλαδή, συμμετοχή των media αλλά και όλων των εργαλείων που ήδη διαθέτουμε. Θα κλείσω λέγοντας πως αυτή η διαδικασία που θα κλείσει με αυτή την έκθεση έχει ένα στόχο. Να αποσαφηνίσουμε πως εδώ δεν μιλάμε για ένα κενό γράμμα το οποίο έχει σκοπό να εξευμενήσει ή να διασκεδάσει τους πολίτες οι οποίοι με τον τρόπο αυτό θα στείλουν απόψεις και τα λοιπά. Όχι. Δεν είναι ένα κέλυφος, είναι μια διαδικασία πολιτικού διαλόγου η οποία είναι πραγματική. Γι' αυτό χρειάζεται ο Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς να δεσμευθεί και αυτός υπέρ αυτών των δράσεων. Ευχαριστώ θέλουμε να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση γιατί τρέχει ο χρόνος και αυτό λόγω των συντονιστών που σας αφήσαν έξω να περιμένετε και ζητώ πάλι συγγνώμη. Ποιος θέλει το λόγο, η κυρία Μίτση. Όπως πολλοί από εσάς σήμερα το πρωί ήμουν στην ακρόαση και ήταν πραγματικά χρήσιμη γιατί ακούσαμε απόψεις από πολλούς. Πολύ χρήσιμες προτάσεις, πολύ χρήσιμες αντιρρήσεις, ενστάσεις και πολύ σημαντικές παρατηρήσεις, τις οποίες πρέπει να έχουμε κατά νου όταν δρομολογούμε μια τέτοια είδους πρωτοβουλία. Θα συμφωνήσω με τόσο είπε μόλις η κυρία Μπεσέρα. Και ως κοιόδης, παρόλο που η γνωμοδότηση ακόμα δεν έχει, η έκθεση δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί, πιστεύω πως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι πολίτες που έχουν λάβει ένα δικαίωμα θα έχουν δικαίωμα και να το εξασκήσουν. Γιατί άλλο να δίνει κανείς δικαιώματα και άλλο να τα εφαρμόζει στην πράξη. Δεν είναι μία απλή ακαδημαϊκή προσπάθεια για να αποδείξουμε ότι εμείς κάνουμε κάτι για τους συμπολίτες μας. Όχι. Πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη. Πρέπει να μπορούν ε, και να τους εκπαιδεύσουμε για να γνωρίζουν πώς υπάρχει αυτό και πώς θα χρησιμοποιηθεί. Είναι πολύ σημαντική η κατάρτιση και η εκπαίδευση, η επιμόρφωση των πολιτών. Να υπάρχουν λοιπόν επαρκείς πληροφορίες σε όλα τα κρατημέλη και εύκολη πρόσβαση σε αυτές για να γνωρίζουν όλοι πώς λειτουργεί το σύστημα. Γιατί το 1 εκατομμύριο υπογραφές, αν είσαι πολίτης και συμφωνείς και δεν ξέρεις πώς μπορείς να συνεισφέρεις σε αυτές τις ε, υπογραφές, ουσιαστικά είναι μία αντίφαση που κάνει την όλη προσπάθεια περιττή. Which will make it easy for, for the the Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως αυτό δεν απευθύνεται μόνο στα, στις ομάδες που κάνουν lobbying. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι πως είναι οι μεμονωμένοι πολίτες που θέλουν κάτι να μας πούν, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό θα αφήσουν να ακουστεί η φωνή τους. Όχι μόνο αυτοί που κάνουν λόμπι, γιατί αυτοί ξέρουν πώς να κινηθούν. Χρειάζεται λοιπόν να αφαιρέσουμε όσο δυνατόν περισσότερους φραγμούς και εμπόδια από όλη τη διαδικασία για να μπορούν οι πολίτες να τη χρησιμοποιήσουν. Όχι μόνο λοιπόν για όσο παίζουν στις επαγγελματικές ομάδες, πραγματική επιμόρφωση έτσι ώστε να τα καταφέρουν όλοι. Ως σκιώδης είμαι έτοιμη να εργαστώ όσο χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε πως οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο δημοκρατίας στο μέγιστο. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιστροφή στη Μάλτα. Τώρα η κυρία με έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω στη γλώσσα μου αυτή τη φορά, Ολλανδικά. Ε, είμαι λίγο απογοητευμένη από την πρωτοβουλία των πολιτών. Όχι από τις προσπάθειες που κάνουν οι πολίτες, αυτές είναι αξιέπαινες, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν τεχνικά προσκόμματα, ε, προβλήματα διάφορα, τα οποία ε, τελικά ε, σταματούν την διαδικασία αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε από τα, μαθήματα, από τα παθήματά μας ε, και τα μαθήματα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Θεωρώ ότι η Επιτροπή ε, πολύ συχνά ε, δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της, το αντίθετο. Πολύ συχνά λέει δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την πρωτοβουλία κτλ. Αλλά όταν εμείς βλέπουμε ε, την πρωτοβουλία πολιτών, ας πούμε, για το TTIP, βλέπουμε ότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν υπογράψει, 300 ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν εμπλακεί. Και το να λέει η Κομισιόν δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, θεωρώ ότι είναι λίγο πολύ εύκολη απάντηση το γεγονός ότι ας πούμε δεν συμπεριλαμβάνεται σε αρμοδιότητές μας σε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό απέναντι στους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε προσοχή στους πολίτες αυτούς και να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ Ήθελα να πω ότι η πρωινή συζήτηση ήταν εξαιρετική, ενδεχομένως η πιο, πιο, το πιο ενδιαφέρον hearing, η πιο ενδιαφέρουσα ε, ακρόαση που ε, άκουσα από τα ήμουν στο Κοινοβούλιο. Πολλές πληροφορίες, πολλοί κόσμος, πολύ ενδιαφέρον γενικά το όλο εγχείρημα. Πιστεύω ότι θα πρέπει στην έκθεση να γίνει αναφορά ε, στο αποτέλεσμα αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας πολιτών ε, να γίνει αναφορά δηλαδή στην ανάγκη συγκεκριμένη ε, δράσης σε μια προηγούμενη ζωή πριν εκλεγώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα συμμετάσχει στην διαδικασία υποβολής αναφοράς ε, και είναι πολλή δουλειά, πολλή προετοιμασία και πραγματικά είναι πολύ αγχωτικό τελικά το αποτέλεσμα να μην είναι ε, το επιθυμητό όταν έχεις περάσει από ένα σωρό δυσκολίες και τεχνικά εμπόδια ε, θέλεις να προχωρήσεις και αυτό που είπε προηγουμένως ενιαία μέθοδος νομίζω μαθηματική νομίζω ότι με βρίσκει σύμφωνη. πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε ξανά λίγο το ε, πεδίο εφαρμογής ε, των ε, πρωτοβουλειών των πολιτών. Ο ορισμός της νομικής πράξης τελικά σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει ας πούμε πρωτοβουλίες πολιτών για θέματα εμπορικά. Ε, ε, και το είδαμε στην περίπτωση της συμφωνίας TTIP δεν έγινε δεκτή η πρωτοβουλία ε, πολιτών και ενδεχομένως νομικά να έχει έρισμα αυτή η θέση αλλά πολιτικά όμως είναι δύσκολο να το δεχτούμε. Επομένως θα πρέπει να δούμε και να αναρωτηθούμε ε, το θέμα της αξιοπιστίας υπάρχουν πολλά ε, τμήματα της πολιτικής τα οποία λόγω των κανόνων μένουν απ' έξω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα πράγμα μόνο θέλω να πω. σήμερα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα. Ακούσαμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απόψεις. Όμως εγώ θέλω να δω τι λένε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί το επιχείρημά μας είναι σαφές τώρα. Ε, το έχουμε βάλει στο τραπέζι. Τώρα αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς ε, ε, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Μπορεί δηλαδή να έχει καλή συνέχεια, μπορεί όμως και να σταματήσει εδώ. Και νομίζω ότι ε, στο σημείο τούτο είναι πολύ σημαντική και μεγάλη η δικιά μας η ευθύνη, έτσι ώστε να μην σταματήσει το θέμα. Εγώ είμαι στους κοιόδες εισηγητές και λέω και επαναλαμβάνω ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να απλουστευθεί ε, και έχουμε μια καλή ευκαιρία εδώ να συνεργαστούμε μεταξύ των συναδέλφων έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε αυτήν την πρόθεση θα πρέπει οπωσδήποτε να μας στηρίξουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να, προχωρήσουν, να προωθήσουν σωστά το θέμα ε, γιατί με τον τρόπο αυτό θα αναπτερωθεί και η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, τώρα έχει κλείσει ο κατάλογος των αγορητών. Μην σηκώνετε πια το χέρι σα να σας πω πώς θα προχωρήσουμε και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Συζήτηση στις 16 Απριλίου. Προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών 31 ε, Απριλίου ε, και ενδεχομένως την Ολομέλεια τον Ιούνιο. anyway, it's far away till the... Βέβαια μέχρι τον Ιούνιο έχουμε καιρό. Το επόμενο θέμα είναι η γνωμοδότηση ε, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών ε, για το νερό. Είσαστε εδώ. Ε, είχαμε φοβηθεί κάποια στιγμή ότι θα είσαστε στο αεροπλάνο αυτή την ώρα. Ευτυχώς είσαστε εδώ. Ναι, ναι, θεώρησα, λέει η ε, κυρία Ούκεν, ότι έπρεπε οπωσδήποτε να είμαι εδώ, έπρεπε να είμαι εδώ, να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Ε, δεν είχα ετοιμάσει κάτι μέχρι να παρακολουθήσω και την ακρόαση σήμερα το πρωί και μπορώ εν συντομία να πω το εξής. Εάν αυτό το εργαλείο της πρωτοβουλίας των πολιτών γίνει σεβαστό, για το καλό των πολιτών και αν θέλουμε να το κάνουμε ε, σεβαστό, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ε, ζητήσουμε την Κομισιόν να καλύπτει και τα υπεσχημένα. Το κάνει μέχρι τώρα γενικά. Είχαμε και την ακρόαση για το δικαίωμα της πρόσβασης στο νερό από μια, ένα χρόνο. 17 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή ΕΝΒΗ με ε, τον πρόεδρο της δικής μας Επιτροπής. Και μάλλον όχι στις 19 Μαρτίου είχαμε ανακοίνωση της Κομισιόν και εκεί ε, μας υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν κάτι. Και μετά όμως τίποτα. Το έρευος δεν έκαναν τίποτα. Ε, φαίνεται ότι έχουν την άποψη ότι καλά τώρα αυτά τα περιβαλλοντικά δεν είναι και για μας τους σπουδαίους ανθρώπους, είναι για πολύ άλλους ε, πολίτες. Ε, αυτή την εντύπωση είχα και με τις πλαστικές μου τσάντες. Αυτό το θέμα που μου είναι τόσο προσφυλές και είχα την εντύπωση ότι το θεωρούν όλοι δευτερεύουσα σημασία. Πιστεύω ότι και στη νέα επιτροπή θα έχουμε την ίδια ε, αντιμετώπιση. Όμως, όμως λέω, εάν λειτουργήσει καλά το εργαλείο αυτό ε, και εάν τώρα έχουμε πλέον κάποιες υποσχέσεις ότι θα το αντιμετωπίσουν θετικά και με σοβαρότητα, ε, να το προωθήσουμε για να, γίνουν, να έχουμε πραγματικά επιτεύγματα. Και εδώ θα μπορούσα να πω επίσης ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία θα είναι καλή και ότι η αναθεώρηση της νομοθεσίας για το νερό θα γίνει με σωστό τρόπο. Αυτό βεβαίως ε, είναι ζήτημα πρωτίστως ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, της ΕΝΒΗ. Εμείς ε, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τα εξής η χρήση της ε, σύμβασης ε, του ε, νερού θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερη, να βελτιωθεί. Δηλαδή πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν ξέρουν ότι μπορούν να προωθήσουν τα αιτήματά τους ενώπιον της δικαιοσύνης, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για τέτοια θέματα. Επίσης η Κομισιόν λέει ότι όλες ε, οι πληροφορίες ε, ε, σχετικά με το νερό και την πρόσβαση στο νερό και τις δυνατότητες κτλ. Όλες οι πληροφορίες, λέω, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους πολίτες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και αν τα υπεσχημένα δεν γίνονται σεβαστά, τότε το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Θα ζητήσω από τους συναδέλφους, ε, τους εσκιώδεις εισηγητές, να πούνε αν έχουν καμιά καλή ιδέα για να ε, την συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μου, ε, να υποβάλουν αυτές τις ιδέες τους μέχρι τη Δευτέρα. Σας καλώ λοιπόν να μου υποβάλετε τις ιδέες σας. Σας ευχαριστώ που είσαστε που δείξατε υπομονή, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα θέματα ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Τα είδαμε και το πρωί και είναι πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάργκρετ. Τώρα δώσω το λόγο στον κύριο Νάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, θα ήθελα και εγώ και από τη σκοπιά της πολιτικής μου ομάδας να δω το θέμα αυτό από πολύ κοντά. Ε, εγώ έχω διατελέσει υπουργός ε, περιβάλλοντος ε, και είμαι και μέλος στην ΕΝΔΙ και επομένως το θέμα της διαχείρισης των υδάτων είναι κάτι που μου είναι ιδιαίτερος προσφυλές. Χαίρομαι που υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία και που εστέφθη από επιτυχία. Δυστυχώς όμως βλέπουμε τώρα ότι η Κομισιόν δεν κάνει και πολλά πράγματα. Μάλιστα μπορώ να πω ότι τα προβλήματα από τη μία πλευρά είναι πολιτικά, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και νομικής φύσεως. Και τελικά δεν ε, προχωράμε και πολύ και δεν μπορούμε να δούμε ε, καθαρά το μέλλον που θα έχει αυτή η ε, πρωτοβουλία ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα για το μέλλον της Ευρώπης και αν εδώ αποτύχουμε θα είναι ένα χτύπημα μοιραίο στην αξιοπιστία μας. Εμείς ε, κάποια στιγμή πήραμε την απόφαση για την πρωτοβουλία των πολιτών γιατί ακριβώς θέλαμε να, να, προκαλέσουμε έτσι έναν ενθουσιασμό στους πολίτες για την Ευρώπη, να τους δώσουμε το λόγο. Εάν δεν έχουν αυτήν την πρωτοβουλία οι πολίτες δεν θα είναι καθόλου ευχαριστημένοι και μάλιστα θα απογοητευτούν όχι μόνο με την πρωτοβουλία αλλά και σε σχέση με την πρωτοβουλία, αλλά θα απομακρυνθούν ακόμα περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την συλλογή των στοιχείων. Και κάτι άλλο που προκύπτει. Γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα γραφείο, μία υπηρεσία ε, που να δίνει πληροφορίες ε, στους ε, πολίτες. Στις 27 περιπτώσεις κατάφεραν οι πολίτες να συλλέξουν πάρα πολλές υπογραφές αλλά τελικά δεν έγιναν, δεκτές, ε, ε, δεν έγιναν δεκτά τα αιτήματά τους ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτά που κάνουμε για την ώρα είναι λίγα. Οι πρωτοβουλίες για το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να ενεργήσουμε με τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μία ατμόσφαιρα συνεργασίας ε, και αυτό θα μπορούσε να γίνει εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέγραφε στην ημερήσια διάταξή του τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δηλώνει την πρόθεσή του, να δηλώνει την θέση του ε, σε αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον που έχουν μαζευτεί πολλές υπογραφές ακόμα και αν το θέμα δεν αφορά αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα προσεγγίσουμε περισσότερο τους ε, πολίτες και εκείνοι με τη σειρά τους θα έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και λέω ότι σε περίπτωση που δεν έχει αρμοδιότητα ε, η Κομισιόν θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να ε, ζητήσει να μετακυλιστούν οι αρμοδιότητες στις χώρες μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης 17 Μαρτίου. Δεν θα είναι όμω τότε μαζί μα, η Μάργκρετ. Θα την αντικαταστήσει κάποιο άλλο από του Πρασίνους. Προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών 27 Μαρτίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μα θα λάβει χώρα στι 5 Μαου. Τώρα, έχουμε μία άλλη γνωμοδότηση για την ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγήτρια τη Σολεδά Καμπεθόνου Ρίφ στην οποία και θα δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Και γιατί έχουμε ένα αντατικό διάλογο, αλλά και γιατί θέλουμε να ακούσουμε στη συνέχεια και κάποιους αναφέροντες. Παρ' όλα αυτά, καταρχάς πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι πρόκειται για μια αρκετά σημαντική έκθεση, διότι αντιμετωπίζει την καρδιά ε, το βασικό νόημα ε, της Ευρώπης σήμερα. Πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε δηλαδή την Ευρώπη, θεμελιώδη δικαιώματα που είναι και η βάση ε, της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Πρόκειται για εκατομμύρια άτομα. Οι διάφορες συνθήκες έχουν ενισχύσει αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οι νομικές αυτές πράξεις συνεχώς. Όλοι ζήσαμε σίγουρα μια κατάσταση που μας ε, δοκίμασε, όπως η οικονομική κατάσταση, η κρίση, οι οικονομικές δυσχέρειες που ήταν σημαντικές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Γι' αυτό και είναι σημαντικό, έχοντας αυτές τις εμπειρίες και αυτά τα βιώματα, να δούμε πώς έχει εξασφαλιστεί προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να δούμε και αν χρειάζεται αναθεώρηση των νομικών πράξεων, αν δεν εφαρμόζονται, αν δεν γίνονται σεβαστά όλα αυτά τα θεμελή δικαιώματα. Θέλω επίση να τονίσω το ότι είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να δουλεύουμε ε, στο μέτωπο τη ε, μη διακριτική μεταχείρισης ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό για οποιοδήποτε λόγο. Ζητούμε λοιπόν και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο η οδηγία που έχει μπλοκαριστεί για την μη διακριτική μεταχείριση, έχει μπλοκαριστεί σε επίπεδο κομισιών να απεμπλακεί η διαδικασία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, για μια κοινωνική Ευρώπη, Ευρώπη των δικαιωμάτων που θα μας διαφοροποιεί από τον άλλο κόσμο, επειδή ακριβώ θα εγγυόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια για όλους, παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουν μεταξύ τους. Τέλος, ένα ζήτημα που τους μήνες αυτούς μπήκε στο προσκήνιο, όπως πάνω χάρη είναι οι αγώνες κατά της τρομοκρατίας, είναι ένα λεπτό ζήτημα αυτό και πολλές φορές ε, έχουμε διάσταση συμφερόντων, διαφορετικές απόψεις ε, και διαφορετικές ευαισθησίες. Κάποιες φορές ε, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση ή οριακά να θεωρηθεί παραβίαση των δικαιωμάτων και όλα αυτά πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά. Είμαι στη διάθεσή σα για να συστήσουμε οποιαδήποτε από αυτέ τι πτυχέ ή οποιαδήποτε άλλη ενδιαφέρει οποιαδήποτε πολιτική ομάδα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε το λόγο. Δεν ήθελα να τοποθετηθεί από ό,τι ξέρω. Άρα. Α, και κανεί άλλο δεν θέλει το λόγο. Άρα θα έχουμε την προθεσμία κατάσταση τροπολογία. Όχι. Α, η Ελεονόρα θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Συγγνώμη, είχα αφαιρεθεί, Πρόεδρε. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την συνάδελφο για την εργασία της, αλλά θα ήθελα να θίξω και κάποια ερωτήματα για να μπορέσουμε να υποβάλουμε ένα, μια γνωμοδότηση η οποία θα βοηθήσει πραγματικά την, ΛΥΜΠΕ, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα πρέπει να καταφέρουμε να αναφέρουμε ε, τις, να αναφερθούμε μάλλον ε, στις συγκεκριμένες αναφορές τις οποίες δεχόμαστε και επί των οποίων όλοι δουλεύουμε. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες σκέψεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναφορές φτάνουν στην Επιτροπή μας και υπογραμμίζουν διαρκώς και όλο και περισσότερο την μεγάλη σημασία που δίνουν οι πολίτες ε, ε, στην, ε, στο προστασία του περιβάλλοντος και στο συνδεδεμένο θέμα της υγείας και που είναι θέματα άλλωστε που αναφέρονται και στη θήκη λειτουργίας στο, στο άρθρο 191 αλλά και για το περιβάλλον και συγγνώμη χάρτες θεμελιωδών δικαιωμάτων και στο 107 άρθρο για την η πρόσβαση στην ε, υγεία, όλα αυτά ε, θα πρέπει να τα δούμε από πάρα πολύ κοντά. Βλέπουμε ότι έχουμε 68 ε, αιτήματα τα οποία σχετίζονται με το ίδιο θέμα. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι θα πρέπει να καλύψουμε επίσης και τα κενά τα οποία υπάρχουν σε ορισμένες ε, ε, χώρες, ε, στις χώρες δηλαδή αυτές οι οποίες δεν έχουν εθνικές επιτροπές αναφορών στις οποίες πρωτογενώς μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες. το θέμα το, της αντιμετώπισης των ε, ανηλίκων και των απαγωγών ανηλίκων είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο με ιδιαίτερη σοβαρότητα θα πρέπει να, αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και σημαντική ευκαιρία ε, για να καταφέρουμε να ε, συλλέξουμε υλικό από τις ε, αναφορές οι οποίες μας φτάνουν και έτσι ώστε να κάνουμε σωστή δουλειά και εδώ και στην Επιτροπή Λίμπε. Ευχαριστώ. Okay, very good. Πάρα πολύ καλά μα τα είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιο άλλο όχι. Να μην επαναλάβω αυτά που είπα για το χρονοδιάγραμμα για να, και να περάσω. Κυρία Ντανόκα, Ντανόκα, θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σκιώδης. Για το ζήτημα αυτό. Είναι πολύ καλή η πρόταση και η συντάκτρια της φωνομοδότησης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτό που ιδίω ε, θέλω να επισημάνω είναι κάτι πολύ θετικό που είπατε, ε, που λέτε στο εισαγωγικό τμήμα Β για τις αναφορές που έχουμε λάβει και οι οποίες έχουν αντικείμενο παραβιάσεις, τις υποθέμες παραβιάσεις, καζόμενες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παραβιάζουν το χάρτη. Αναφέρεστε στο άρθρο 51 του χάρτη. Όμως, αυτό που είναι σημαντικό και δεν αναφέρεται εδώ, είναι ότι ακριβώς το άρθρο 51 ε, δεν μας επιτρέπει να αναλάβουμε δράση όταν λαμβάνουμε τέτοιες είδους αναφορές. Η Κομισιόν επανειλημμένως μας λέει ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμβει. Γιατί το άρθρο 51 λέει ότι μπορούμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές μόνο, κάποιες απόψεις. Υπάρχουν όμως διασυνοριακές ε, περιπτώσεις, αρπαγές παιδιών και άλλα προβλήματα με παραβιάσεις ανθρωπίνων θεμελιωδών μάλλον δικαιωμάτων. Η Κομισιόν όμως συνήθως λέει ότι όχι, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πολύ θα ήθελα λοιπόν η γνωμοδότηση αυτή να εστιάσει πιο πολύ στα θέματα αρμοδιότητα, ειδικότητα, αν μπορώ να το πω έτσι, τη δική μα επιτροπή και οι τροπολίε που θα καταθέσουμε να καταδεικνύουν αυτά τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την εφαρμογή του χάρτη και την εξέταση συγκεκριμένων αναφορών. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής, σωστής εφαρμογής του χάρτη. Πρέπει δηλαδή ναι, κάποιε αναφορές μπορούμε να τι κρατήσουμε ανοιχτέ και να ασκήσουμε κάποια πολιτική επιρροή ή να τις κλείσουμε. Αλλά τίποτε περισσότερο, ακριβώς λόγω του άρθρου 51. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ υποθέτω ότι και αυτή θα έχει να πει κάτι σχετικά. Απλά σας κάνω την πρόταση αυτή. Να αναφέρουμε και εμείς τα συγκεκριμένα προβλήματα της Επιτροπής Αναφορών όταν έχουμε να κάνουμε με αναφορές ε, στο χάρτη των κοινωνικών δικαιωμάτων. Πρόεδρος, τώρα που άκουσε τη συντάκτη γνωμοδότηση και τη σκιώδη εισηγήτρια η Κομισιόν ε, εξακολουθεί να μην θέλει να λάβει το λόγο ή άλλαξε άποψη. Yes. Thank you. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Φοβούμαι ότι την ίδια απάντηση ακριβώς θα λάβετε. Αυτή που έχετε ακούσει τόσο συχνά. Γνωρίζω Γνωρίζω ότι ο χάρτης των λοιπόν θεμελιωτών δικαιωμάτων πρίμα φάκε όταν το πορτακούει κανείς ε, μπορεί να φαντάζεται κανείς ότι περιλαμβάνει τα πάντα αλλά το άρθρο 51 ξεκαθαρίζει ότι είναι εφαρμοστέο για τα θεσμικά όργανα και κατά δεύτερον για τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν όταν εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι δεν σας ικανοποιεί καθόλου αυτό ε, ως Επιτροπή Αναφορών. Είναι όμως πολιτικό το ζήτημα, είναι πολιτικό πρόβλημα και αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε και να επιβεβαιώσουμε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Okay. And the Χρονοδιάγραμμα. 16 Μαρτίου, 6 το απόγευμα, λίγη προθεσμία κατάσταση τροπολογιών. 16 Μαρτίου. Κοντά είναι αυτή η ημερομηνία. Θα ψηφίσουμε στις 16 Απριλίου στην Επιτροπή μας και μάλλον ή τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο στην Ολομέλεια, αλλά δεν είμαστε ακόμη σίγουροι. Αυτό λοιπόν είναι το χρονοδιάγραμμα. Και τώρα κυρίε και κύριοι, προσδεθείτε παρακαλώ, διότι έχουμε να συζητήσουμε ένα ακόμη θέμα και αυτό είναι οι αναφορές για συζήτηση Επιτροπή επί τη βάση, μάλλον είναι η γνωμοδότηση σχετικά με τι συστάσει προ την Επιτροπή όσον αφορά τι διαπραγματεύσει για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, το λεγόμενο που Ο κ. Βαλέ, εισηγητή μα, παίρνει μέσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ξεκινήσω, θα θέλω να υπογραμμίσω πω κατά την προετοιμασία αυτή τη γνωμοδότηση προσπάθησα να συμπεριλάβω όσο το δυνατόν περισσότερε απόψει και αναφορέ οι οποίε ελήφθησαν υπόψη. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γραμματεία για την καταπληκτική δουλειά που έχει κάνει για να πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αναφορές το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε οι συνόψεις να είναι έτοιμες το συντομότερο δυνατόν. Ξέρετε πως η που αποτελεί ένα από τα μεγάλα θέματα στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκαλεί μεγάλες και έντονες συζητήσεις σε επίπεδο ενδιαφερομένων. Οι πολίτες μας εξέφρασαν πάρα πολλές ανησυχίες, τις οποίες στη δική μας Επιτροπή χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Και τα θέματα αυτά μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες. Σχετίζονται με την ποιότητα των εισαγωγών τροφίμων, με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών για την ψηφιακή αυτοδιάθεση, τη διαφάνεια, τα θέματα οικονομικού αντικτύπου και την προστασία των επενδυτών στα πλαίσια του μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Κατά τη συνεδρίαση του Μαρτίου θα συζητήσουμε αυτά, αυτές τις αναφορές και εγώ πρότεινα στους συντονιστές να επιλέξουμε τις αναφορές βασιζόμενοι στα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Αυτό θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και παράλληλα έστειλα και μία σύσταση, έστειλα μάλλον σε αυτούς και τις συστάσεις και να τονίσω εδώ πως για κάθε θέμα ε, έχουν ε, και όλα μου τα επιχειρήματα. Στη συνάντηση που έκανα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου είπαν πως θα κάνω ό,τι μπορούν για να είμαστε έτοιμοι για το Μάρτιο με τις απαντήσεις για τις συγκεκριμένες αυτές αναφορές. Ελπίζω πως θα μας πούν περισσότερα για την απόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις συστάσεις μου, για την δημόσια διαβούλευση και τα όσα έχει πει και ζητήσει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που η δική μας Επιτροπή αποφάσισε να ετοιμάσει αυτή τη γνωμοδότηση, γιατί αποδεικνύει πως είμαστε δεσμισμένοι προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσοι με βοήθησαν και να πω πως η γνωμοδότηση αυτή θα είναι πολύ επιβοηθητική για τις επόμενες γνωμοδοτήσεις και αναφορές που θα λάβουμε για την TTIP οι οποίες ε, θα μπουν και αυτές στα σκαριά όσο περνάει ο χρόνος. Εν πάση περιπτώσει ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Σκιώδης και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Πείτε μου πως, ε, μάλλον ε, θυμηθείτε πως αυτή είναι μια μη νομοθετική πρόταση, οπότε πρέπει να είναι λιγότερο από μια σελίδα. Μην το ξεχνάτε. Thank you very much. πρώτα απ' όλα, κυρία το λόγο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Γιαροσλάβ, γιατί το σχέδιο αυτό γνωμοδότησε για την επόμενη συνάντησή μας ε, το Μάρτιο ε, θα μας βοηθήσει να προλάβουμε το πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα ε, για την ψηφοφορία της ΣΥΝΤΑ και την Ολομέλεια και για να καταφέρουμε όσοι ανησυχούν να λάβουν μια απάντηση ακόμα και αν αυτό σημάνει πως η διαδικασία θα επιμηκυνθεί γιατί θα φτάσουν σε μας και άλλες αναφορές ε, σύντο χρόνο και θα πρέπει να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλων αυτών των όγκων αναφορών. Ένα-δύο θέματα έχω, τα οποία δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς από τη γνωμοδότηση και για να σας ε, πω περίπου τι τροπολογίες θα υποβάλουμε. Ξέρω πως η δική μας εντολή είναι να καλύψουμε τις αναφορές οι οποίες καταφτάνουν, αλλά ένας μεγάλος αριθμός ε, καλύπτουν το μηχανισμό διακανονισμού για διαφορές ε, σε περίπτωση επενδύσεων και δεν μπορούμε αυτό να το αφήσουμε γιατί εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση και αυτή η διαβούλευση ε, γίνεται τον ίδιο χρόνο μαζί με κάποιες από αυτές τις αναφορές. Δηλαδή με τη στιγμή που υποβλήθηκαν αυτές οι αναφορές. Αυτό πρέπει να το αναφέρουμε στη γνωμοδότηση. Και θα πρέπει επίσης να κάνουμε κάποιες σκέψεις για το τι είπε αυτή η διαβούλευση όπου το 97% των όσων απάντησαν, 150.000 απαντήσεις ήταν η μεγαλύτερη ε, τέτοια προσπάθεια που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν απολύτως αρνητικές. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη εμείς αυτή τη μαζική απόκριση των συμπολιτών μας. Άρα λοιπόν και τις διαβουλές για το θέμα του μηχανισμού θα πρέπει να τις συμπεριλάβουμε. Λυπάμαι κάπως που δεν ε, ασχοληθήκαμε με το γεγονός πως προσπάθησε να ξεκινήσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την TTIP και αυτή η πρωτοβουλία αποκλείστηκε επειδή δεν βασιζόταν σε νομική πράξη, αλλά σε προσωρινό έγγραφο που ήταν η διαπραγματευτική εντολή. Νομίζω πως ως Επιτροπή εμείς εδώ μπορούμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Είναι κομμάτι του ε, πεδίου αρμοδιοτήτων μας και όλα αυτά αποδεικνύουν πως υπάρχει πάρα πολλή ανησυχία για την TTIP. Οι πολίτες δηλαδή έχουν θίξει πάρα πολλέ ανησυχίες, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των όσων λαμβάνουμε. Είναι θέματα τα οποία μας αναφέρουν οι πολίτες. Ξέρω πως όλοι βιαζόμαστε. Υπάρχει το θέμα της διαφάνειας. Σε κάποιο σημείο μιλάμε για το πώς χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει τη διαφάνεια και μιλάμε για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Θα πρέπει επίσης να δούμε και κάποιες από τις επικριτικές σκέψεις που έχουν ακουστεί για το reading room, δηλαδή για τα έγγραφα τα οποία θα μπορούσαν να θεωρούνται δημόσια, βρίσκονται σε μια αίθουσα στην οποία δεν μπορούν να μπουν οι ευρωβουλευτές, δεν μπορούν να μπουν οι πολίτες, σε, μια, σε ένα αναγνωστήριο δηλαδή, όπου δεν μπορούμε να μάθουμε εμείς το περιεχόμενο αυτό και να δούμε τι έχει πει και ο διαμεσολαβητής για αυτά. μια και υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες σχετικές στις αναφορές που λαμβάνουν. Περιμένω λοιπόν τα, όσα θα πούμε το Μάρτιο και θέλω να δω τι συνέχεια θα δοθεί. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ούκεν έχει το λόγο. Πολλοί από εσά δεν θα είναι στις 17 Μαρτίου είναι κατά το ίμιση τυρκουάζ εβδομάδα. Εγώ θα πάω στην Παλαιστίνη με την αντιπροσωπεία. Και ξέρω πως δεν θα έχουμε και όλες τις τροπολογίες, όλες τις γλώσσες μέχρι τότε. Οπότε ας βρούμε έναν τρόπο να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Σας προειδοποιώ ότι είναι πολύ σημαντική η συνάντηση του Μαρτίου για τη δική σου έκθεση για Αροσλάβ, όπου πέφτει την αρχή μιας εβδομάδας ε, της ΚΟΑΣ και λυπάμαι πάρα πολύ που συμβαίνει αυτό. Το θέμα αυτό θα πρέπει να το δούμε με πολύ προσοχή. Πάρα πολλές αναφορές έχουν φτάσει και μπορεί στο μέλλον να δούμε η δική μας νομοθεσία να υποσκάπτεται ακόμα και αν μας δηλώνουν τώρα πως αυτό δεν θα συμβεί. Υπάρχουν τόσα πολλά που διακυβεύονται και να σας πω πως πέρσι όταν τελειώσαμε ήμουνα πολύ ικανοποιημένη από την διαφάνεια που είχαμε πετύχει ε, με το φαρμακευτικό κλάδο για τις ε, νοσοκομιακές δοκιμές και νομίζω ότι οι πολίτες καλωσορίζουν αυτή τη διαφάνεια και τελικά λίγο μετά ξαφνικά μπήκε στον ε, πάγο αυτή η, η οδηγία από τον αντίστοιχο κλάδο στην Αμερική. Είπαν πως αυτή είναι από την νομοθεσία που θέλουμε να καταργηθεί. Και αυτό μας λένε τώρα και οι φαρμακοβιομηχανίες στην Ευρώπη. Θέλουν όλη αυτή τη διαφάνεια να την καταργήσουν για την οποία εμείς δώσαμε μάχες. Και συμφωνείς μεν μαζί μας, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίζεις πως υπάρχει πραγματικά κίνδυνος και δεν ξέρουμε αν όντως θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Αυτές οι δηλώσεις ότι θα δημιουργήσει πάρα πολλές θέσεις εργασίας είναι πολύ αμφισβητήσιμες. Και το γεγονός πως δεν θα έχουμε τελωνία κτλ. Μα τι σημαίνει αυτό, έτσι κι αλλιώς ε, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο βάρος από τα τελωνία μεταξύ μας. Είμαι υπέρ, ε, είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Αλλά εδώ δεν έχει να κάνει με το ελεύθερο εμπόριο. Έχει να κάνει με το πώς θα εναρμονίσει κανείς. Και εκεί θα πρέπει στη διαδικασία μέσα να εξασφαλίσουμε που θα κάνουμε συνειδητά βήματα. Όπως είπαμε και για το μηχανισμό τον ίδιο. Δηλαδή εμείς παραμερίζουμε τα δικά μας δικαστήρια και δημιουργούμε ένα εργαλείο το οποίο έχει να που σχετίζεται με το εμπόριο με χώρες που έχουν πολύ αδύναμα νομικά συστήματα. Και αυτό θα ισχύσει μεταξύ ΕΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, ας πούμε πως η κατάσταση είναι πολύ πιο δραματική από ό,τι έχουμε δηλώσει δεν είναι μόνο το ελεύθερο εμπόριο, είναι και το πώς εμείς θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Γι' αυτό το λέω, είμαι πολύ τρομαγμένη και σίγουρα θα δούμε πολλά και ίσως μάλιστα παγιδευτούμε. Πάντως ευχαριστώ για την, την έκθεσή σου και την ευγένειά σου. Και σε προειδοποιώ, θα χειροτερεύσει η κατάσταση, θα πάρεις πολύ περισσότερες αναφορές. Δεν μοιάζεις τροπαγμένος, Γιάροσλαβ. Α, όχι, μόνο τον θυμώνω πραγματικά, τον τρομάζω. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Η κυρία Αλβιόλ Γκουσμάν. Ευχαριστώ. Η Γκούε, λαμβάνοντας υπόψη πως αυτή η Επιτροπή πρέπει να ασχολείται με τη διαφάνεια, το δικαιωμένο μέρος των πολιτών, την εμπλοκή των πολιτών και δεδομένων, του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι διαπραγματεύσεις, Πιστεύουμε πως η γνωμοδότηση δική μας θα πρέπει να είναι φιλόδοξη και πραγματικά κρίσιμη και επικριτική. Από τις 560 συνεδρίσεις ε, που έγιναν για τη συμφωνία αυτή, το 92% έγινε με τους ενδιαφερόμενους και τα λόμπι και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και ελάχιστε συνεδρίσεις έγιναν με κοινωνικά κοινωνήματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και συνδικάτα. Καταλαβαίνω πως η γνωμοδότηση θα πρέπει να, ε, να παρουσιάζει πως κρύβονται πληροφορίες από ε, το κοινό. Ούτε εμείς οι βουλευτές δεν έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες και στο αναγνωστήριο το οποίο υπάρχει για να μπορέσουμε να διαβάζουμε τα έγγραφα δεν μπορούμε να μπούμε όλοι και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε την επιστολή ε, αυτό που έκανε ο αρχηγός των διαπραγματεύσεων των, Ευρωπαϊκών, των Ευρωπαίων διαπραγματευτών στον ε, ομόλογο του στη ΣΥΠΟ, όπου είπαν πως τα έγγραφα της διαπραγμάτευσης θα κλείσουν, θα είναι απόρριτα για το κοινό για 30 χρόνια. Μα, μιλάμε τώρα για σκοταδισμό. Ε, οι συστάσεις του διαμεσολαβητή, της διαμεσολαβήτρες μάλλον, για το πώς θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, που θα είναι τα έγγραφα τα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μας κάλεσε να επιβάλλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτές τις συναντήσεις. Υπόθηκε λοιπόν πως θα πρέπει να ξεκινήσει μία διαβούλευση 150.000 άτομα πήραν μέρος στη διαβούλευση Κομισιόν και 97% είπαν όχι στο μηχανισμό αυτό που επιτρέπει στους πολυεθνικές να ε, ε, καταστρατηγήσουν τους κανόνες της δικής μας δημοκρατίας και θα πρέπει στη γνωμοδότηση αυτό να φαίνεται, όπως επίσης και μια κριτική πιο βαθιά προς τη συνθήκη αυτή που θα επηρεάσει όλους τους κλάδους ζωής μας, κρατικές υπηρεσίες, τρόφιμα, απασχόληση, γεωργία, εργασιακά δικαιώματα, πρόσβαση στα φάρμακα, στις πληροφορίες, με πολύ αρνητικό τρόπο. Να πούμε λοιπόν πως θα εργαστούμε για το θέμα αυτό και θα υποβάλουμε τροπολογίες κτλ. Ευχαριστώ. That's good. Πολύ ωραία. Η Ελεονόρα τώρα έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την, για την εργασία του. Θα ήθελα ε, να κάνω κάποιες νέες σκέψεις ε, χωρίς να χρειαστεί να ε, επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν συνάδελφοι και με τα οποία συμφωνώ. Μια και εκπροσωπούμε εδώ την Επιτροπή <clears throat> Αναφορών, θα πρέπει να δούμε πώς σχετίζεται το θέμα αυτό με τη δουλειά μας. Ε, και ε, μπορούμε να διαπιστώσουμε λοιπόν ότι ο προβληματισμός που εκφράζεται από τους πολίτες μέσω των αναφορών ε, αφορά κυρίως ε, την αμφισβήτηση της ε, αλήθειας των λεγόμενων όσον αφορά τις εμπορικές επαφές, το περιβάλλον, την υγεία και κυρίως την αηφορία αυτής της και την βιωσιμότητα αυτής της συμφωνίας. νομίζω ότι η Επιτροπή μας είναι το καλύτερο φόρουμ, το ιδεώδες φόρουμ έτσι ώστε να γίνει η ανταλλαγή απόψεων με τους πολίτες ε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αδιαφάνειες ε, και ε, άλλωστε το είπε και η Σανεφός δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε να μην μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο reading room. Δεν μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε τις επιπτώσεις αυτής της συνθήκης και για τις δύο υπήρους. και η αρχή της ε, ε, πρόληψης ε, είναι μια βασική αρχή η οποία αφορά και τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και θα πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί σε αυτή τη συνθήκη έτσι ώστε η εργασία να είναι σωστή. Κατά τα λοιπά βεβαίως χαίρομαι πολύ που με τη διαδικασία του κατεπήγοντος θα ασχοληθούμε με αυτές τις αναφορές. Ανυπομονώ. Πολύ ωραία. Η Κομισιόν θέλει να πάρει το λόγο και να μας δώσει, να μας κάνει κάποια σύντομα σχόλια. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για οικονομία χρόνου δεν θα αντιδράσω σε κάθε ένα σχόλιο ξεχωριστά. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά και για την Επιτροπή σας εδώ και για την συζήτηση της 17ης Μαρτίου. Πρώτον, γνωρίζετε ότι η συμφωνία TTIP είναι ένα από τα κυριότερα ζητήματα της Επιτροπής που αντιμετωπίσουν οι συναδελφοί σας στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Πολλά από τα ζητήματα τα οποία γίνεται σήμερα έχουν ήδη φυγεί στα πλαίσια της ε, ΙΝΤΕ. Και ήδη στις 17 Μαρτίου μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά ε, σε αυτά τα οποία ε, τα στοιχεία της συμφωνίας τα οποία αφορούν το εμπόριο. Δεύτερον, σε μερικές περιπτώσεις στην συζήτηση που γίνεται, ε, στην δημόσια συζήτηση, δημιουργείται η εντύπωση ότι η κοινή γνώμη είναι κατά του TTIP εμείς ε, όμως κάναμε μια σφιγμομέτρηση και τη γνωρίζουμε τη σφιγμομέτρηση αυτή η οποία δείχνει ότι αντιθέτως η πλειοψηφία είναι υπέρ καταρχήν μια συμφωνίας. Από την ε, οπτική γωνιά της ε, Κομισιόν είπαμε και βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε κάποιους προβληματισμούς, ε, πολλοί εκ των οποίων αναφέρονται ε, και αναφέρθηκαν σήμερα στην ε, Επιτροπή, να γίνουν οι διασαφηνίσεις οι οποίες δεν έχουν γίνει ακόμα. Εν συντομία να πω δύο λόγια για την διαφάνεια, μια και είναι ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Juncker ε, έχει θεσπίσει την διαφάνεια σαν μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές της. Στις 25 Νοεμβρίου η Κομισιόν ενέκρινε ανακοίνωση με συγκεκριμένη αναφορά στο TTIP. Δεν θα τη διαβάσω και δεν θα επαναλάβω όλες τις λεπτομέρειες που εκεί περιέχονται. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι έχουμε ήδη αρχίσει να ε, εφαρμόζουμε αυτήν την χωρίς προηγούμενο και σημαντική πρωτοβουλία για την ε, διαφάνεια μπορείτε να βρείτε ένα σωρό κείμενα και πληροφορίες ε, στο ίντερνετ για όλα τα ζητήματα τα οποία συζητούνται ε, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών. Μπορείτε να δείτε ακριβώς ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ως διαπραγματευόμενου μέρους. Στο διαδίκτυο λοιπόν και στους ιστοτόπους που είναι διαθέσιμοι μπορείτε να βρείτε ένα σωρό χρήσιμες πληροφορίες για τους γύρους των συζητήσεων, για τα διάφορα ζητήματα, τα διάφορα στοιχεία τα οποία συζητιούνται και εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε σχετίζεται με την ουσία των διαπραγματεύσεων. Έχουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα πολύ συγκεκριμένο και λεπτομερές σύστημα το οποίο ήδη εφαρμόζεται έτσι ώστε να μπορούμε να πιάσουμε το σφιγμό του πολίτη και να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Νομίζω ότι για πολλές από τις ε, σε πολλές από τις υπηρεσίες της Κομισιόν ε, είναι κυρίαρχο ζήτημα αυτό της ε, επαφής με τους πολίτες, ε, της επικοινωνίας με τους πολίτες. Ας πούμε, στη διάρκεια κάθε γύρου συζητήσεων έχουμε μία συγκεκριμένη συνάντηση των εμπλεκομένων μερών, συνεδρίαση η οποία ή μπορεί να την παρακολουθήσουν όλοι στο διαδίκτυο, είναι web streamed because the standards were uh, mentioned here, was uh, a question or a fear. Υπάρχει και πολλή φόβος ή ανησυχία γιατί μπορεί κάποιοι να φοβούνται πως για τα χημικά για παράδειγμα θα μειωθούν τα επίπεδα προστασίας και εμείς έχουμε οργανώσει πολλές δημόσιες συναντήσεις με τους εμπλεκομένους για να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες της ίδιας της πρότασης Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε αν όντως αληθεύει, αν όντως υπάρχει λόγος ανησυχίας. Βεβαίως δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε στον κόσμο τι θα σκέφτεται, αλλά είναι πρώτον σημαντικό να δώσουμε τις φοβερίε και δεύτερον να εξηγήσουμε τι ακριβώς διαπραγματευόμαστε. Έχουμε μια συμβουλευτική ε, ομάδα για την TTIP, έχουμε πολλές δράσεις εξωστρέφειας προς τους πολίτες. Εγώ προσωπικά Πολύ συχνά πηγαίνω στη Γερμανία, την πατρίδα μου και πηγαίνω σε διαλόγους με τους πολίτες για την TTIP. Οπότε αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε πάρα πολλούς πόρους γιατί για μας είναι προτεραιότητα. Για να εξηγήσουμε στους πολίτες τι ακριβώς κάνουμε. Γιατί πιστεύουμε πως αυτό συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση και για ποιο λόγο υπάρχουν ανησυχίες να τις δούμε μία-μία, να δούμε τους φόβους και μία τελευταία παρατήρηση Είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Αυτή τη στιγμή ε, ετοιμάζεται και η τελική μορφή της έκθεσης του Διαμεσολαβητή που θα δημοσιευθεί και πρέπει να σας πω πως γενικά ο θεσμός αυτός αυτή τη στιγμή πενεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προσπάθειες που γίνονται. Η διαμεσολαβήτρια μίλησε για, όλα, για πολλά θέματα τα οποία εξετάσαμε όλα. Κάποιες από τις παρατηρήσεις που έκανε τις εφαρμόσαμε, άλλες τις σκεφτόμαστε. Και ίσως αυτό είναι κάποια από τα ζητήματα που θα μπορούσαμε σε μια επόμενη συνεδρίαση, για παράδειγμα 17 Μαρτία, να συζητήσουμε. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθώ σε όλα αυτά τα σημεία. Ευχαριστώ πολύ που τα είπατε τόσο λεπτοπεριακά και σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο ανοιχτός και πρόθυμος να μπείτε σε, αυτή την, σε αυτό το συνεχιζόμενο διάλογο με την Επιτροπή μας και με άλλες επιτροπές. Τώρα λοιπόν το χρονοδιάγραμμα είναι το σχέδιο 17 Μαρτίου, προθεσμία για τροπολογίες 23 Μαρτίου και ψηφοφορία 16 Απριλίου. Έτσι θα προχωρήσουμε. Γιάρικ, τα εξήγησες καλά, δεν θα σου ξαναδώσω το λόγο. Τα πούμε αργότερα, γιατί τώρα πια έφτασε η ώρα να προχωρήσουμε. Να δώσουμε το λόγο δηλαδή στους αναφέροντες οι οποίοι βρίσκονται εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα γιατί πρέπει να μάθουμε περισσότερα για τα όσα συμβαίνουν. Με ιδιαίτερη χαρά θα καλέσω στην συνεδρίαση αυτή την κυρία Μπεατρίς Γκαρότ την κυρία Κριστίνα Μαρσίγιας και από την αντιπροσωπεία της κοινότητας της Βαλένσια την κυρία Παλάου Ταρέγα όπως επίσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε κάποιους εκπροσώπους. Θα δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ένα βίντεο. Ξέρετε ποιο είναι το υπόβαθρο, είναι το ατύχημα που έγινε στο μετρό της Βαλένσια που έχασαν τη ζωή του 43 άτομα και άλλοι 47 τραυματίστηκαν. Τώρα λοιπόν θα δούμε το βίντεο και μετά θα του ακούσουμε. Hm.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 ¿Puedo hablar? να μιλήσω. En las imágenes acaban de ver, στις εικόνες που μόλις είδατε φαίνεται ποια ήταν ε, η στάση της ε, κυβέρνησης Βαλένθια και του, της διεύθυνσης του μετρό σε μια τραγωδία πραγματική ε, χειραγωγήθηκε η κοινοβουλευτική έρευνα, δεν υπήρξε διαφάνεια για το ατύχημα, ε, λογοκρίθηκαν δε και τα δημόσια μέσα επικοινωνία. 43 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 46 τραυματίστηκαν. Οι νεκροί ε, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι ανεπίστρεπτο. Δεν κλείνουν οι πληγές αυτές. Η μόνη τέτοια, για μετά από τη τραγωδία, η μόνη αν θέλετε παρηγοριά, είναι να αληθούν τα αίτια της τραγωδίας και να λαμβάνονται μέτρα για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ωστόσο, η δράση της ε, βαλυνθιανής κυβέρνηση ήταν το αντίθετο ακριβώς, ψεύδι και χειραγώγηση. Εμείς θύματα αυτής της τραγωδίας δεν το αξίζαμε αυτό. Και καμία κοινωνία δεν ε, αξίζει πολίτες οι οποίοι είναι γατζωμένοι στην εξουσία σε κόστος και σε βάρος των πολιτών που τους έχουν ε, εκλέξει να τους υποστηρίζουν. Δημιουργήσαμε την Ένωση των Θεμάτων του Μετρό. Θέλουμε να αγωνιστούμε για τα θεμελιώδη μα δικαιώματα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ε, από το 2006 εργαζόμαστε και προσπαθούμε να αλλάξουμε ε, και αντί για σιωπή να έχουμε απαντήσει, αντί για τιμωρησία να έχουμε υπευθυνότητα, ευθύνη και αντί για έλλειψη σεβασμού να έχουμε αξιοπρέπεια. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια μετά από αυτή την τραγωδία δεν ε, πρέπει ε, να φανεί ε, ότι αυτό που θέλουν να συγκαλύψουν τελικά είναι ότι δεν υπήρχε ασφάλεια τη μέρα του ατυχήματο. Έχουμε μιλήσει με δικηγόρου, με ακτιβιστέ, τον των πολιτών, με συνδρομικού υπαλλήλου, με ανώνυμου πολίτε μας έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και σιγά σιγά καταφέραμε πολλές πληροφορίες να τις βγάλουμε στο φως και να ε, δείξουμε ότι είναι ψέματα αυτά τα οποία έλεγε η κυβέρνηση και το μεγαλύτερο επίτευγμά μας πέρυσι ήταν όταν καταθέσαμε αυτή την αναφορά και ξεκίνησε εκ νέου η δικαστική έρευνα, η δικαστική διερεύνηση στην Βαλένθια και έχουμε και τρεις που κατηγορούνται για ελλείψεις ε, στην ασφάλεια. Θέλουμε να πούμε ότι ε, ουσιαστικά ε, τις ε, πληγές μας μετράμε εδώ. Έχουν χαθεί άτομα την οδύνη και την οδύνη μας, την αγανάκτησή μας απέναντι στην ανυμποριά που νιώθαμε γιατί η κυβέρνηση είχε τηρήσει αυτή τη στάση. Σε αυτά όλα αντιπαραβάλαμε την αποφασιστικότητά μας για τον αγώνα. Μετά το 2006 Έχουμε καταλάβει ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στου πολιτικού να συνεχίζουν να ψεύδονται για να παραμείνουν στην εξουσία. Πρέπει να λάβουμε τι ευθύνε των πράξεών του. Και αυτό δεν πρέπει να του το εμποδίσει το γεγονό ότι έχουν την απόλυτη πλειοψηφία. Εμείς δεν ζητούμε τόσα πολλά. Αυτό που ζητούμε είναι απλά ε, κάτι που θα κάνει την κοινωνία να βελτιωθεί που θα προσπαθήσει να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια στις αστικές μεταφορές. Γι' αυτό πολλές φορές ζητήσαμε από την βαλαθιανή κυβέρνηση να ε, τηρεί την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν το έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Επίσης σημαντικό θεωρούμε είναι ένα που ε, από τα σημεία της αναφοράς να εγγυαόμαστε την πολυμορφία και την αμεροληψία στις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει ένα κανονισμό για τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ σχετικώ. Και στόχο μα είναι η αναζήτηση τη δικαιοσύνη. Κάτι που δεν το βρήκαμε στη χώρα μα, γι' αυτό και ήρθαμε στις Βρυξέλλες. Για μα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρη σημερινή, διότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση θα κάτσει και θα αναλύσει τι καταγγελίε μα τα αιτήματά μα. Για πρώτη φορά εδώ στις Βρυξέλλες θα αναζητηθούν ευθύνε για τη διαχείριση του ατυχήματο. Ελπίζουμε να μα στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα παρακαλώ, μη μας αντιαψεύσετε τις ελπίδε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Κριστίνα Μαρσίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε γιατί μας δώσατε την ε, δυνατότητα ε, να έρθουμε εδώ ε, αποδεκόμενοι την δικιά μας Ετη ε, τη δικιά μας αναφορά όσον αφορά αυτό το ατύχημα ε, στην ε, Βαλένθια και επίσης να σας ευχαριστήσουμε γιατί έχετε ήδη μοιράσει και τα έγγραφα τα οποία έχουμε φέρει στα μέλη της Επιτροπής. Μοιραζόμαστε βεβαίως την οδύνη και τον πόνο μαζί με, όλους, όλα τα θύματα αυτού του ατυχήματος και θέλουμε οπωσδήποτε να διευκλευκανθούν τα αίτια. Την ίδια μέρα που ε, συνέβη το, το, συμβάν, ε, ήδη άνοιξε η ε, δικαστική έρευνα, η οποία όμως το 2008 αρχιοθέτησε την υπόθεση λέγοντας ότι απλώς υπήρχε μια υπέρβαση ταχύτητα. και ε, γι' αυτό έγινε ο εκτροχιασμό 80 χιλιόμετρα την ώρα αντί 40 που ήταν το επιτρεπτό όριο. Ε, εμείς ε, όμως ζητήσαμε να ξαναανοίξει το θέμα μετά από την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Τον μήνα Φεβρουάριο μάλιστα έχει υποβληθεί ένα, μια έκθεση από εμπειρογνώμονα τον οποίο είχε ορίσει η δικαστική αρχή ε, ε, όπου αναφέρεται ότι το τρένο δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, ε, το πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στην κυκλοφορία. Δεν είναι δυνατόν τα χρήματα και η οικονομική αποζημίωση να πάρει την θέση ενός αγαπημένου ε, ανθρώπου που χάθηκε. Αλλά παρόλα αυτά θεωρούμε ότι οι ε, αρχές, ε, η κυβέρνηση της Βαλένθια θα πρέπει να δείξει την ε, ε, τη θέση της όσον αφορά ε, αυτό το ατύχημα. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει και σε πολιτικό επίπεδο να αναζητηθούν οι ευθύνες ανάλογα με την εκπροσώπηση που υπάρχει στο Κοινοβούλιο γιατί ούτως ή άλλως πλειοψηφικά ελαμβάνονται οι αποφάσεις και ούτως ή άλλως και το χρονοδιάγραμμα της Ερευνητικής Επιτροπής έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την ε, Βουλή της Μπαλένθιας. Ε, ε, Η λειτουργία της Επιτροπής ήταν αυτή που έπρεπε να είναι και και στις 48 υποθέσεις οι οποίες μελετήθηκαν σε κάθε περίπτωση ελήφθησαν οι αποφάσεις κατά πλειοψηφία και σε όλες τις ε, περιπτώσεις και από διάφορες πολιτικές ομάδες ε, επιβεβαιώθηκαν αυτά. Επίσης ε, εμφανίστηκαν ενώπιον της Βουλής τα 32, 32 άτομα τα οποία απήντησαν στις ερωτήσεις που ελεύθερα υπέβαλαν τα μέλη όλες ε, οι πληροφορίες ε, που είχε η διοίκηση ε, δόθηκαν στα δικαστήρια και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Ούτε οι μηνυτήριες αρχές ούτε η υπεράσπιση παραπονέθηκε για μη πρόσβαση σε τέτοια έγγραφα το σύστημα αυτόματης πέδησης της γραμμής, των τρένων της γραμμής 1 θεωρήθηκε ε, κατάλληλο ανάλογα με, την, ε, ε, με τα στοιχεία τα οποία παρουσίαζε και τις ιδιαιτερότητες της γραμμής αυτής. Δεν διαφαίνεται από την μελέτη της Επιτροπής, της Επιτροπής η οποία μελέτησε το θέμα από την εταιρεία ότι θα έπρεπε να υπάρχει αλλαγή, ότι ε, συγγνώμη, η αλλαγή του συστήματος από ΦΑΠΣΕ ε, ΑΤΠ ε, προκάλεσε οποιοδήποτε πρόβλημα. Ε, και άλλωστε στην Επιτροπή Ασφάλειας ε, της Κυκλοφορίας ε, τον Σεπτέμβρη του 2005 αναφέρεται σαφώς το θέμα αυτό και μάλιστα η, κανένας από τους δύο συνδικαλιστικούς εκπροσώπους δεν είχε ζητήσει αντικατάσταση του συστήματος βράχη ή μακροπρόθεσμα. Ε, δεν ε, προκύπτει επίσης ότι ε, πριν από το ατύχημα του 2006 είχε συμβεί άλλο παρόμοιο ατύχημα στην ίδια στροφή στροφή από την οποία περνάνε κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο και πάνω τρένα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουμε εδώ ότι σε αυτή τη στροφή δεν έχει ξαναγίνει ατύχημα, έχει γίνει σε άλλο σειρμό του ιδίου τρένου. Ε, και επίσης ε, στην γραμμή αυτή ε, λαμβάνονται υπόψη και καταγράφονται μάλλον αναλυτικά όλα τα ατυχήματα και όλα τα συμβάντα τα οποία μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της διαδρομής των τρένων. Παρόλα αυτά το σύστημα ε, ε, το, το σύστημα το οποίο λειτουργεί, στο, του οποίου λειτουργούν ε, τα τρένα και το, το σύστημα των πελμάτων των τρένων έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι το σωστό. Επίσης, όσον αφορά την κάλυψη από πλευράς του σταθμού της, του, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης της Βαλένθια, ε, τις τρεις πρώτες μέρες ε, μετά από το ατύχημα ε, είχαμε περισσότερες από 30 ώρες καταγεγραμμένες πληροφόρησης, καταγεγραμμένες στα αρχεία της ραδιοτηλεόρασης της, Βανίας, της Βαλένθια. Όσον αφορά τώρα την παραβίαση των ε, ε, ε, ευρωπαϊκών νομοθεσιών πρέπει να πούμε ότι μετά από σχετική ανάλυση δεν, δεν διαπιστώνεται αυτό το οποίο υπονοεί η οργάνωση ότι δηλαδή υπάρχει παραβίαση του άρθρου 2 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον πολιτικό πλουραλισμό και όσον αφορά την δημοκρατική αντιπροσωπευτικότητα από νομικής ε, πλευράς ε, το, η χάρτα θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων εφαρμόζεται μονάχα ως δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όσον αφορά τώρα θέματα ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην προκείμενη περίπτωση. Πάντως, ανεξάρτητα από το εάν και κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, οπωσδήποτε πρέπει να πούμε ότι στην προκείμενη περίπτωση υπήρξε απόλυτη διαφάνεια και ελευθερία έκφρασης ε, ε, όσον αφορά όλες τις βαθμίδες της νομικής αντιμετώπισης του, του θέματος. Γενικώ πρέπει να σας πω ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι στη διάθεσή σας να σας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα όσα συζητάτε, σχετικά με αυτές τις ε, Ευχαριστώ πολύ. Γιορτάνο Βίγκο, παρακαλώ, από την Κομισιόν. Grazie, signora Presidente. Ε, a Για να σας πω ειλικρινά δεν έχω και πολλά να προσθέσω γιατί τα περισσότερα έχουν ήδη υποθεί. Όσον αφορά ε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία για θέματα συνδροδρομικών μεταφορών, όντως αυτή δεν εφαρμόζεται στις τοπικές μεταφορές και στις μητροπολιτικές μεταφορές. Θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές δεν ενδείκνυται ε, αυτή η νομοθεσία για τοπικές ε, ε, συγκοινωνίες. Αυτό βεβαίως δεν εμποδίζει τις εθνικές ή τοπικές αρχές να εμπνευστούν από την Ευρωπαϊκή ε, Οδηγία ε, την στιγμή που καθορίζουν τους κατάλληλους κανόνες ε, για τις τοπικές συγκοινωνίες ή μεταφορές. Βεβαίως ε, δεν μπορούν να αντιγραφούν ακριβώς ε, οι ίδιες τεχνικές ε, διαλειτουργικότητας γιατί βεβαίως για τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τις μετροπολιτικές και αστικές συγκοινωνίες οι, οι, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι οι ίδιες. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρεται εδώ, ε, στην αναφορά αυτή, και που μελετάτε ήδη από τις ε, Ισπανικές Αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπισμένη ότι οι Ισπανικές Αρχές ε, το συντομότερο δυνατόν θα παράσχουν όλες τις απαραίτητες και σημαντικές πληροφορίες στη διάρκεια των διαφόρων διαδικασιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα ιδιαίτερα προσφυλές θέμα, γι' αυτό λοιπόν θέλω και εγώ να μιλήσω στη δικιά μου γλώσσα. Κύριε Βαλέσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βράτω με τις ευκαιρίες για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Και τώρα θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστούν με σεβασμό οι οικογένειες αυτές και να λάβουν όλη την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη από την εθνική και την περιφερειακή κυβέρνηση της χώρας τους. Αλλά νομίζω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε σε κάπως δύσκολη θέση, από την έννοια Ακούσαμε για το τέτοιο σιδηροδρομικό πακέτο από την Κομισιόν που εγκρίθηκε πριν από δύο χρόνια. Από αυτό εξαιρείται το τραμ το μετρό και τα τρόλεϊ ε, από το πεδίο της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους επικουρικότητας. Ως Επιτροπή Αναφορά φυσικά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τις οικογένειες των θυμάτων και τα θύματα να βρουν δικαίωση, αλλά πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ περιορισμένα. Διότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας το νομικό πλαίσιο και την αρχή της επικουρικότητας. Thank you, Mrs. Albiol. Ευχαριστώ, Αλβιόλ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω την ε, Βαλενθιανή Ένωση των Θυμάτων του Μετρό, τη αναφέρουσε που είναι ένα παράδειγμα αξιοπρέπεια και αγώνα για μα. Ε, να πω απ' την άλλη ότι είναι λυπηρό που χρειάστηκε να έρθουν εδώ να διεκδικήσουν κάτι που του αρνήθηκε η κυβέρνηση τη Βαλένθια, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια δηλαδή και έπρεπε να έρθουν στι Βρυξέλλε για να ακουστεί φωνή του σε κοινοβούλιο. Αυτό το δυστύχημα είναι το πιο ε, ζωφερό επεισόδιο ε, στην ιστορία τη Βαλένθια και από τι πιο δραματικέ σελίδε τη ε, Ισπανική και Ευρωπαϊκή Ιστορία δεν ανελήφθησαν πολιτικές ευθύνες. Διότι, όπως υπόθηκε, κάθε μέρα στην πλατεία της Βίρχεν Ντεβαλέθια ε, και το λέμε κάθε, σε κάθε επέτειο 3 Ιουλίου είχαμε 43 νεκρούς και 46 τραυματίες αυτό το δυστύχημα. Το λιγότερο που θα μπορούσαμε ε, να περιέχουμε ήταν ε, αυτή η γλώσσα που χρησιμοποίησε ε, πρόσωπος του ε, Κόμματος. Μέσα σε πέντε μέρες, ούτε καν σε ένα μήνα, ξεκαθάρισαν το θέμα, τους αρνήθηκαν έγγραφα, μαρτυρίες, καταθέσεις και είδαμε και πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και στο βίντεο. Επίσης ε, έκρυψαν ε, παλαιότερα ατυχήματα και ποτέ ε, δεν είδαμε και το ημερολόγιο συντήρησης ή βλαβών και ζημιών. Εμείς θέλουμε να γίνει σεβαστή πολιτική πολυμορφία, πλουραλισμός. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια τώρα της εκπροσώπου της Βαλενθιανής Κυβέρνησης, που δυστυχώς είναι το πρόσωπο μιας κυβέρνησης και την υποστηρίζει ενώ δεν θα έπρεπε, υπήρξε χειραγώγηση, υπήρξε λογοκρισία και όπως είπε και αναφέρουσα παραβιάζεται ε, το άρθρο 11 για την ελευθερία έκφρασης, ε, το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Καλό θα ήταν να υπάρξει αποστολή ευρωβουλευτών ε, που θα μεταβεί επιτόπου για να διαλευκάνει το τι έγινε, να μιλήσει με τους ερευνητές, με τους πρώην εργαζόμενους ε, του τύπου που του ζητήθηκε να καλύψουν ε, τα γεγονότα και να μιλήσουμε και με εμπειρογνώμονε. να δούμε τι μέτρα ε, ασφάλειας αστόχησαν και με αυτό το αυτόματο σύστημα πέδηση, τι έγινε και κυρίω, βέβαια για να μην ξανασυμβεί ποτέ ένα τέτοιο δυστύχημα στο μέλλον. Dear colleagues, we are running short. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, δύο ακόμα λεπτά. Θα ήθελα να ζητήσω από τους διερμηνείς ε, εάν συμφωνούν να μας ε, δώσουν ακόμα 10 λεπτά. Δεν βλέπω. Πέντε λεπτά δίνουν οι διερμηνείς. Εντάξει, πέντε λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο μακρύς κατάλογος Ισπανών συναδέλφων ε, δεν θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο. θα δώσω τον λόγο στην κυρία Εστάρας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε και προηγουμένως, εμείς ε, βεβαίως ε, δίνουμε τη στήριξή μας προς όλα τα θύματα και τους 43 νεκρούς και τους 47 <clears throat> τραυματίες που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ από τις οργανώσεις. Ε, και η οργάνωση των ε, άκουσα προσεκτικά και τις δύο παρεμβάσεις ε, και πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση της Βαλένθια με τη δέουσα επιμέλεια και άμεσα με ταχύτητα ε, ε, αντιμετώπισε. Ε, δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνουμε υπόψη τους ανεξάρτητους πραγματογνώμονες που όλοι κατέληξαν στο ότι υπήρχε υπέρβαση του ορίου ταχύτητος που ήταν 40 χιλιόμετρα εκεί ενώ το τρένο έτρεχε με 80 χιλιόμετρα. Δεν έχουν καταγραφεί προηγούμενα παρόμοια ατυχήματα στον ίδιο σειρμό. Ε, επίσης η Πολυτεχνική Σχολή της ε, Βαλένθια, της Βαρκελόνης και άλλης ε, μίας πόλης κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα. Στην τελευταία έρευνα η οποία άνοιξε πρόσφατα έχουμε μια καινούρια επιτροπή πραγματογνωμόνων και πρέπει να πω ότι όποιος και αν ε, κυβερνάει οι ε, ε, διερευνητικές επιτροπές λειτουργούν πάντοτε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών ομάδων, υπάρχει πλουραλισμός κτλ. Το σημαντικό ούτως ή άλλως δεν είναι η Επιτροπή Διερεύνησης, είναι η νομική ε, Επιτροπή, δηλαδή η νομική ανεξάρτητη διερεύνηση η νομικη ανεξαρτητη διαρευνηση η οποια θα καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχουμε 306 αρχεία τα οποία αναφέρονται στη γραμμή 1 ε, και 30 και πλέον ώρες μετάδοσης ε, προγραμμάτων τις τρεις πρώτες μέρες του ατυχήματος. Ε, κοιτάξτε τώρα, εάν ε, ε, ο τρόπος με τον οποίο έγινε, τα ωράρια μετάδοσης και τα λοιπά μπορεί να μην μας ικανοποιούν, αλλά παρόλα αυτά οι ίδιοι οι τεχνικοί οι οποίοι εκλήθησαν να να ε, ε, ε, μιλήσουν στην Επιτροπή και στην, στην Επιτροπή Έρευνας και στην αστυνομία και στο δικαστήριο είπαν ότι ήταν ελεύθεροι, ότι δεν είχαν κανένα περιορισμό στον τρόπο με τον οποίο θα μετέριδαν το θέμα. Εν πάση περιπτώσει τώρα έχει ξανανοίξει το θέμα, θα, θα προχωρήσει, θα φτάσει μέχρι το τέρμα του. και πιστεύω ότι τα όσα έκανε η κυβέρνηση μέχρι τώρα ήταν σωστά, η τοπική κυβέρνηση, θα προχωρήσει το θέμα, θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά ε, και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουμε προσωπικά, ε, συγγνώμη, προσεκτικά τα όσα λένε τα εμπλεκόμενα μέρη. Uh, one more speaker and that will be... Εντάξει, ακόμα έναν μπορώ να... Η κυρία Σεμπάγιος. Ακόμα ένας ομιλητής. Porque... Sí, quedan cinco minutos. Put it If Κοιτάξτε, εάν θέλετε να μιλήσετε αγγλικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά οι διερμηνείς μας έχουν δώσει δύο... Εγώ είχα ζητήσει, για το, είχα ζητήσει το λόγο προηγουμένως και πραγματικά ήθελα να μιλήσω σε αυτή την επιτροπή. Εγώ ήθελα απλώς να πω ε, ε, να αναφερθώ σε κάτι που είπα η εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Βαλένθιας ότι δεν υπήρξε καμία ε, επικάλυψη. Ναι, αλλά αν δεν είχε υπάρξει καμία επικάλυψη, καμία απόκρυψη, τότε δεν θα είμαστε εδώ σήμερα με κάθε αν, αν είχε γίνει σε βάθος διερεύνηση χωρίς, με πλήρη διαφάνεια δεν θα είμαστε σήμερα εδώ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 δεν είσαστε ε, οι ε, επόμενοι. Ο κύριος Μάχιο έχει ζητήσει πρώτα το λόγο, έχει καταγραφεί πολύ γρήγορα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να, να εκφράσω τη στήριξή μου σε όλες τις οικογένειες ε, και στους, προς τους εκπροσώπους των θυμάτων. Ακόμα και ένα θύμα να αντιπροσώπευαν, εγώ θα τους σεβόμουν το ίδιο, όχι τόσους που εκπροσωπούν. Εγώ είμαι εδώ και πολλά χρόνια μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, αναρωτιέμαι γιατί μέχρι τώρα δεν έφτασε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα μέχρι τώρα ε, στην Επιτροπή Αναφορών που συζητάμε τόσα πολλά σημαντικά θέματα. Ε, κοιτάξτε, Προφανώ ε, δεν έφτασε μέχρι εδώ γιατί ε, δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι παρεβιάζεται οποιαδήποτε ε, ενωσιακή νομοθεσία. Εν πάση περιπτώσει, πολλά υπόθηκαν, πολλά ακούσαμε. Πιστεύω ότι πολλά είναι απολύτως άδικα και άλλα σωστά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το σημαντικό τώρα είναι να αναλάβουμε δράση. Ε, δεν, ε, έχει, ε, δεν έχει έννοια τώρα να συζητάμε για τις πολιτικές αυτές ομάδες, τα πολιτικά αυτά κόμματα τα οποία εγχειρηματοποίησαν αυτό το θέμα για τις πολιτικές τους εκστρατείες. Νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρόμαστε αυτή τη στιγμή που έφτασε εδώ η αναφορά και ότι μέσω της μελέτης της θα έρθουν οποιασδήποτε επιφυλάξεις και νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και να προχωρήσει. Okay, we will lose our interpreters in 30 seconds. Σε 30 δευτερόλεπτα δεν θα έχουμε άλλο, άλλο τους διερμήσεις στη θέση γι' αυτό σας προτείνω το εξής. Πρώτον, εκ μέρους αυτής της Επιτροπής να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε εσάς που ήρθατε εδώ και μοιραστήκατε την οδύνη, ε, την, ε, τον πόνο σας, ε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε εδώ και τόσο καιρό. Πρόκειται για μια ανθρώπινη τραγωδία. Κατανοούμε τη θέση σας και σίγουρα είμαστε πλήρης συμπάθειας και κατανόησης για το τι έχετε περάσει και τι περνάτε ακόμα. Επειδή αυτή είναι όμως ε, η δεύτερη ε, δικαστική έρευνα και διαδικασία που ξεκινάει, ε, θα παραμείνει ανοιχτή αναφορά και εμείς στην Επιτροπή μας θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την υπόθεση αυτή. Δικαστήριο δεν είμαστε βέβαια, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η μάχη που δίνεται. Ακούσαμε ότι δεν ισχύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στα μέσα ελαφράς τροχιάς. Ε, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λοιπόν εδώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Θα ζητήσω πληροφορίες, θα εξεταστεί η υπόθεση. Παρακαλώ να μας διατυπώσετε προτάσεις. Εάν εμείς ως νομοθετική επιτροπή ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι, ε, ενημερώστε μας. Να είστε βέβαιοι όμως ότι είναι κάτι που πραγματικά μας έχει συγκινήσει και μας πείσατε ότι κάτι πρέπει να γίνει και θα το παρακολουθούμε και εμείς ε, του σύνεκες. Λυπούμε πολύ που δεν μπορώ να δώσω ε, τον ε, λόγο σε όλους, γιατί πρέπει όσο είναι διερμηνής να κλείσω την συνεδρίαση αυτή και αν θέλετε μπορείτε να έχετε διμερείς επαφές με τους βουλευτές μας. Ευχαριστώ πολύ. Anyway, would like ε, to, uh, constar in acta que no se me ha dado la palabra, que solo ha dado la palabra. Eh, ήθελα απλώς να καταγραφεί στα πρακτικά ότι δεν, ε, δεν μου δόθηκε ο λόγος, ότι δεν δόθηκε ο λόγος στην ομάδα των ε, σοσιαλιστών ε, και ότι μας βρίσκει απολύτως αντίθετη αυτή, αυτός ο αστείος τρόπος με τον οποίο ε, αντιμετώπισε το θέμα η uh, that in the draft of, the, uh, of this uh, committee